Dear colleagues, Συνάδελφοι, καλώς ήρθατε. Εγκρίνετε την ημερήσια διάταξη. Ωραία, ευχαριστώ. Σύντομες ανακοινώσεις έχουμε. Διόρθωση στην οδηγία για τις πληρωμές διανεμήθηκε στις 9 Μαρτίου. Δεν λάβαμε σχόλια, οπότε προτείνω να υποβάλουμε το κείμενο στην Ολομέλεια σύμφωνα με το άρθρο 131 παράγραφος 2. Και τώρα καλωσορίζω τον Ντανιέλ Νουή, πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στο πλαίσιο του ενιαίου ελεγκτικού μηχανισμού. Έχουμε την ετήσια έκθεση λοιπόν όπως έχουμε συμφωνήσει στη διοργανική συμφωνία μας, η οποία καλύπτει τις εποπτικές δραστηριότητες ε, για το 2017 και έχει ενημερωθεί βεβαίως σύμφωνα με τις ε, πιο πρόσφατες αποφάσεις. Που έχουμε ήδη συζητήσει μεταξύ μας ε, και με τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό το 2017 ήταν ε, το τέταρτο έτος όπου η ΕΚΤ ε, ήταν ο ενιαίος επόπτης ε, της Ευρωζώνης οπότε αναμένουμε να ακούσουμε την κυρία Νιουή για την προόδο της ΕΚΤ, τις δραστηριότητες του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού και τις προτεραιότητες του τραπεζικού τομέα. Όπως ξέρετε, ε, το Κοινοβούλιο ενέκρινε και το σχετικό ψήφισμα την 1η Μαρτίου, όπου παρουσιάσαμε τις ε, θέσεις μας για τα διμερή ζητήματα. Ένα σχετικό θέμα βεβαίως είναι το θέμα των εξυπηρετούμενων δανείων, που όπως ε, ξέρετε αφού τελικά ο ενίος οπτικός μηχανισμός εξέδωσε την τελική εκδοχή της ε, προσθήκης ε, ε, πριν η Κομισιόν παρουσιάσει το σχετικό πακέτο. Υπάρχουν λοιπόν πολλές σχετικές ειδήσει. Και κάποιοι ανησυχούσαν βεβαίως όσον αφορά την προσθήκη ε, αυτή ότι δεν είχε ληφθεί υπόψη η άποψη του Κοινοβουλίου και όπως ξέρετε αν παρακολουθήσει κανείς τις αλλαγές ε, στο Word αντιλαμβάνεται ότι υπήρξαν κάποιες ε, προσπάθειες αλλαγής για τη μη αυτόματη φύση της προσθήκης οποίας καλώς καλωσορίζω. Και βεβαίως Κοινοβούλιο ε, κάναμε μια νομική αξιολόγηση αλλά θα την κάνουν και οι νομικές μας υπηρεσίες και νομίζω ότι μία αυτόματη φύση των ε, εποπτικών προσδοκιών έχει πλέον ανακοινωθεί και θα εστιάσουμε περισσότερο στον ε, διάλογο και θα λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση της κάθε τράπεζας ε, ξεχωριστά. Αυτό είναι κάτι το θετικό. Βέβαια, τώρα έχουμε ένα ζήτημα ε, το οποίο αφορά κάποιες διαφορές μεταξύ των υποπτικών προσδοκιών και του τι έχει προτείνει η Κομισιόν ως πλαίσιο του πυλώνα 1 Οπότε η αξιολόγησή μου για το τι θα ακούσουμε είναι ότι όταν οριστικοποιηθεί πλέον το προληπτικό πλαίσιο του πυλώνα 1, καλό θα είναι να υπάρξει μια ευθυγράμμιση των ρυθμιστικών προσδοκιών με την ομοθεσία χωρίς βεβαίως να επηρεάζεται να επηρεάζονται τα προνόμια εποπτικού μηχανισμού για περαιτέρω απαιτήσει ε, στον πυλώνα 2. Αλλά βεβαίω υπάρχει μια γενικότερη οριζόντια φύση των ε, προσδοκιών ε, για να μην υπάρχει σύγχυση στις τράπεζες για το τι πορεία πρέπει να ακολουθήσουν Δηλαδή αυτή του πυλώνα 1, αυτή του πυλώνα 2, ειδικά αν υπάρχουν μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές. αυτό είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση. Έχουμε χρόνο ακόμα και ακριβώς θα πρέπει να εγκρίνουμε μια νέα νομοθετική πρόταση το συντομότερο δυνατόν για να έχουμε σαφείς κανόνες για τις τράπεζες λαμβάνοντας υπόψη ότι μιλάμε για ένα πακέτο διαφόρων μέτρων που, όπως είπε η Κομισιόν, είναι αναγκαίοι για να λειτουργήσουν. Έχουμε και άλλα ζητήματα, το πρόβλημα με τις τράπεζες της Λετωνίας και το έλλειμμα που υπάρχει αυτή τη στιγμή όσον αφορά το πλαίσιο καταπολέμησης του ξεπλήματος χρήματος και την ομοιογένεια αυτή στο εθνικό επίπεδο. Όλα αυτά θα τα πει φαντάζομαι η κυρία Νουή. Μακρηγόρησα εν πάση περιπτώσει και σας δίνω τον λόγο. Σας ευχαριστώ και καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Με μεγάλη χαρά σας ε, παρουσιάζω την ετήσια έκθεση της ΕΚΤΕ για τις εποπτικές δραστηριότητες. Όπως και τα προηγούμενα χρόνια θα κάνω μια επισκόπηση των βασικών μας δραστηριοτήτων για το 2017 και πολύ συγκεκριμένα θα μιλήσω για τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τη στοχευμένη αναθόρηση ε, των εσωτερικών μοντέλων, Brexit, θεματικές αναθεωρήσεις και διάφορους άλλου θεσμικού φορεί Τέλος, ε, που χρειάζεται να λάβουμε άλλα μέτρα για να ενισχύσουμε την Τραπεζική Ένωση. Θα αρχίσω λοιπόν με μια επισκόπηση των πεπραγμένων για την Τραπεζική Ένωση. Το 2017 ε, το οικονομικό περιβάλλον βελτιώθηκε και ενισχύθηκαν οι κεφαλιακές θέσεις και οι ισολογισμοί των τραπεζών. Βλέπουμε από το τρίτο τρίμηνο του 2016 από 13,7% ε, φτάσαμε στο 14,3% μέσα σε ένα χρόνο. Ε, και με την προσπάθεια που έγινε ε, για τη μείωση των NPLs τα μη εξυπηρετούμενα δανεία μέσα σε ένα χρόνο έπεσαν σε ποσοστό από το 6,5% στο 5,2%. Το 2017, τους πρώτους 9 μήνες, ε, για την ανάκαμψη, για τις, ε, τα, τελειτουργικά κέρδη, επίσης σημειώθηκε μια πολύ σημαντική αύξηση, αλλά μειώθηκε το net interest margin, ε, οδηγώντας μας σε πολύ μεγαλύτερη επιστροφή σε σχέση με τις επενδύσεις, που ανέρχεται σε 7% σε σχέση με το 5,4% το 2016. Έτσι ευθυγραμμίζονται περισσότερο με ε, τους ομοτήμους τους ε, στη ΣΥΠΑ. Γενικότερα ε, υπάρχουν διακυμάνσεις ανάμεσα στις τράπεζες το 2017 επίσης για πρώτη φορά οι άμεσα επιτηρούμενες ε, τράπεζες ε, ε, βγήκαν από την κατηγορία του big to fail και το Εποπτικό Συμβούλιο του ΕΚΤΕ μπόρεσε να συμβάλλει σημαντικά στην αποτροπή των κρίσεων. Θα ήθελα τώρα να περάσω σε λεπτομέρειες για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Ξέρετε ότι αυτό είναι προτεραιότητα για μας και η προσέγγιση μας περιστρέφεται γύρω από τρεις άξονες. Πρώτον, ποιοτική καθοδήγηση προς τις τράπεζες για τα μη εξυπηρετούμενα δημοσίευσαμε σχετικό έγγραφο το Μάρτιο 2017 ε, προϋποθέτει αυτό ότι ε, εκπονούνται φιλόδοξα αλλά και εξόπλες στρατηγικές για τα μη εξυπηρετούμενα οι τράπεζες ε, και εφαρμόζονται σχέδια δράση για την αντοπισή τους. Ε, δεύτερον, εποπτικός διάλογος όπου οι κοινέ εποπτικές ομάδες ε, εκ του παρακολουθούν τις προκλήσεις των τραπεζών και τις στρατηγικές ε, για τα κόκκινα δάνεια. Έχουν ε, αποφέρει ήδη καρπούς ε, οι στρατηγικές. Βλέπουμε ότι έγιναν πολύ σημαντικές προσπάθειες από, μεγάλα, από μεγάλες τράπεζες για μη εξυπηρετούμενα που ανέρχονται σε 200 δις. Παρόλα αυτά, σε πολλά κράτη-μέλη εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα και αυτό αποτρέπει τον δανεισμό και δεν επιτρέπει στις τράπεζες να υποφελήσουν από την οικονομική ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Τρίτο, ε, σχε... Τρίτος άξονας, στις 15 Μαρτίου 2017 δημοσιεύσαμε μετά από δημόσια διαβούλευση ένα έγγραφο. Η, διαβούλευση ήταν από τον Οκτώβριο μέχρι τον Δεκέμβριο και βλέπουμε στο παράδειγμα αυτό το εγγράφο ότι για λόγους διαφάνειας ε, έχουμε συγκεκριμένες προσδοκίες ε, για την τροφοδότηση με νέα μία εξυπηρετούμενα δάνεια ε, και αυτό είναι η βάση του διαλόγου με μεμονωμένες τράπεζες. Αναθεωρήσαμε το παράρτημα υπό το φως των σχολείων που λάβαμε κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης ε, και μεταξύ άλλων λάβαμε υπόψη τις νομικές ανησυχίες που καλύψαμε στη τελευταία ακρόαση τον Νοέμβριο, δηλαδή Θέσαμε ως νέα ε, διορία τον ε, Απρίλιο του 2019 για την αναθεώρηση του συστήματος για τα κόκκινα δάνεια. Σε σχέση με τα backstops για τις ε, προληπτικές εποπτείες σε σχέση δηλαδή με, την, με το χειρισμό των δάνειων που αποδεικνύεται ότι είναι κόκκινα, κάναμε τις προτάσεις μας στο παράρτημα. Πρόκειται για επιπρόσθετες πρωτοβουλίες και από κοινού θα υποστηρίξουμε τις κοινέ προσπάθειες για την μετώπιση αντιμετώπιση των κόκκινων δανείων στο μέλλον. Ε, η στοχευμένη αναθεώρηση τώρα των εσωτερικών μοντέλων, ε, Project TRIM, ε, αυτό διεξάγεται νη συνεργασία με τις Εθνικές Αρμόδιες Αρχές μέχρι το 2019. Βαίνει αισίω το ΤΡΙΜ, ε, περίπου in situ 19 επιθεωρήσεις, έγιναν το 2017 και στο μεταξύ έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα του προγράμματος ΤΡΙΜ, περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο σε σχέση με ζητήματα όπως ε, η διακυβέρνηση του μοντέλου, η επικύρωσή του και μέσα από προληπ εποπτικέ αποφάσει έχουμε ήδη διεκπαιρεώσει αυτά τα ζητήματα. Τώρα, προετοιμασίε για το Brexit. Παρακολουθούμε το του συνεχής ε, το θέμα τη μετεγκατάσταση ε, των τραπεζών και τα σχετικά προγράμματά τους. Ε, βλέπουμε ότι λαμβάνουν αποφάσει για τα σχέδια Brexit και μετεγκαθίστανται στην Ευρωζώνη. Επίσης, νέε πολιτικές ούτως ώστε ε, να είναι κατάλληλα προετοιμασμένε οι τράπεζε για το Brexit και να έχουν τις κατάλληλες δομέ διακυβέρνηση. Επίσης, να είναι ορθή διαχείριση με ένα βιώσιμο business model για τις οντότητες που έχουν μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κοινοποιήσει ποιο χρόνο χρειάζεται για την επεξεργασία των αιτημάτων μετεγκατάσταση και για αυτέ τι τράπεζε που επιθυμούν μετεγκατάσταση ή επέκταση δραστηριοτήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και χρειάζονται αδειοδότηση για την επέκταση των δραστηριοτήτων μετά το Brexit το η έκθεση συνεργασία με τις ε, αρμόδιες εθνικές αρχές αναμένει το ταχύτερο δυνατόν τα αιτήματα, αλλά το αργότερο μέχρι το τέλος του 2018, αν δεν έχουν ήδη υποβληθεί, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την επεξεργασία αυτών των αδειών πριν τον Απρίλιο του 2019, εάν ε, υποβληθούν εκπρόθεσμα. Τώρα, θεματικές αναθεωρήσεις. Ε, πολύ σημαντικό ε, εποπτικό εργαλείο, διότι ε, πρόκειται για την διευκολύνση την επιταχυμένη εποπτική αντίδραση της ΕΚΤΕ και διαπιστώνουμε ότι πρόκειται για μία από τις προτεραιότητες της ΕΚΤΕ για το 2017, δηλαδή αξιολόγηση μεταξύ άλλων το βαθμό στον οποίο οι αρχές είναι προετοιμασμένες για να εφαρμόσουν το IFRS 9 σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων για την αξιολόγηση αντικτύπου για τα προληπτικά αριθμητικά στοιχεία. Επειδή υπάρχουν Ευχαριστώ. Ε, στην κερδοφορία των τραπεζών μεγάλες διακυμάνσεις. Ε, με ιδιαίτερη προσοχή ε, αναλύουμε τα επιχειρησιακά μοντέλα με γνώμονα την κερδοφορία. Και συνεχίζουμε λοιπόν τη θεματική αναθεώρηση, ξαναλέω, για το 2017. Εξετάζω όλο συγκεκριμένα την κερδοφορία και έτσι θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των τραπεζών. Η κοινή εποπτική ομάδα στη συνέχεια θα αναλάβει δράση κατά τράπεζα, ανά τράπεζα. Ε, σε σχέση με τη συνολική διακυβέρνηση ε, την ε, δυνατότητα ομαδοποίησης θα ασχοληθούμε με σύνολα ομάδες τραπεζικών ιδρυμάτων σε περίπτωση που σε περιπτώσεις όπου ε, θέλουμε να αναλάβουμε άμεσα δράση θα το κοινοποιούμε σε αντίστοιχες επιστολές. Για τις, ε, τη συνεργασία με τις εθνικές αρχές τώρα παρακολουθούμε τις ε, περιπτώσεις ε, τραπεζικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης, δηλαδή ανακοινώνουμε την εποπτεία μας με τρόπο που είναι συμβατό με την κουλτούρα τους και ε, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας έχουμε κοινά πρότυπα, που τα έχουμε εφαρμόσει, όμως ε, εμφανίζονται και νέα για την αδειοδότηση λιγότερο ε, σημαντικών ε, τραπεζικών ιδρυμάτων με πρότυπα fintech. Εγκρίναμε νέα μεθοδολογία και εναρμονίσαμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούν τη διακριτική τους ευχέρεια εθνικές αρμόδιες αρχές για λιγότερο σημαντικά τραπεζικά ιδρύματα. Για το 2019 έχουμε τέσσερις Εποπτικέ πρωτοβουλίε ε, Τις τρεις μεταφέραμε από το 2017. Πρώτον, είπαμε, επιχειρησιακά μοντέλα για τους drivers, ε, για τους ε, κινητήριους παράγοντες, δηλαδή τις κερδοφορίες των τραπεζών. Δεύτερον, η έμφαση στα ε, μη εξυπηρετούμενα δάνεια και έκθεση συγκεντρώσεις ε, εκθέσεων και τρίτων στο, στη διαχείριση κινδύνων. Η το τρίμ θα συνεχιστεί, η αναθεώρηση των μοντέλων. Θα συνεχιστεί και η εποπτεία σε σχέση με την αναθεώρηση των ιστορικών διεργασιών των τραπεζών ναι, για τα εργαλεία όπως θα ονομάζουμε ICAP για την ρευστότητα. Στη συνέχεια, υποπτικές δραστηριότητες με πολλαπλές διαστάσεις διαχείρισης σε κινδύνου, όπως παραδείγματο χάρη τα τεστ ε, ε, αντοχής ε, του 2018 για το Brexit. Κλείνοντας, Μία αγνήσια τραπεζική ένωση δεν χρειάζεται μόνο αυτούς τους ε, τρεις επιλώνες, αλλά πρέπει να καταπολεμήσει και τον κατακαιρματισμό και το fencing, ε, την απομόνωση των ε, εθνικών τον κατακαιρματισμό που οφείλεται στο ring fencing, τον αποκλεισμό των εθνικών ε, αγορών. Ε, ε υπάρχουν ναι, ακόμη κολλήματα ε, κανονιστικού χαρακτήρα σε σχέση με τη διακριτική αυχαίρεια που έχουν τα κράτη-μέλη, όπως παράδειγμα χάρη σε σχέση με την αποτροπή μεγάλων ε, βαθμών έκθεσης. Ε, πρέπει να εγκριθεί ε, περαιτέρω νομοθεσία σε σχέση με τις ήδη ισχύουσες οδηγίες για την αξιολόγηση της κερδοφορίας. Επίσης, δημιουργούνται προβλήματα διότι 19 διαφορετικά εθνικά σετ, εθνικές δέσμες νομοθετικών ρυθμίσεων καλείται να εφαρμόσει η ΕΚΤΕ. Για το στο πακέτο Βασιλεία 3 και συμπεριλαμβανομένου και του νέου κανονισμού κανονιστικού ε, πλαισίου για τη διαχείριση του κινδύνου αναμένουμε σημαντικές εξελίξεις ε, και ε, η Κομιτεία της Βασιλείας φυσικά αντιμετωπίζει εμπόδια, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται επιχειρήματα για να επιβραδύνει τη διαδικασία. Χρειάζεται Δικλείδε ασφαλεία σε κανονιστικού χαρακτήρα επαρκή για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Η εναρμόνιση θα πρέπει να συνοδεύεται από μια ολοκλήρωση τη ε, δημοσιονομική αρχιτεκτονική με ένα αξιόπιστο backstop για το SRF, το Κοινό Ταμείο, για να καλύψει τα θέματα φερεγγιότητας ε, και τη στήριξη των τραπεζών ε, σε σχέση και με το ΕΝΤΙΣ φυσικά, την εγγύηση των καταθέσεων. Το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια πρόταση ευθυγραμμίσης του κανονισμού σε σχέση με τις επενδυτικές εταιρείες, ε, με τις διατάξεις για τις τράπεζες, ε, όπως ε, παρακολουθούνται και ελέγχονται από την ΕΚΤ στα πλαίσια της προετοιμασίας του Brexit, διότι αυτές οι επενδυτικές εταιρείες έχουν πάρα πολύ σημαντικές διασυνορικές δραστηριότητες και θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο λαμβάνουμε τα απαιτούμενα μέτρα, ούτω ώστε οι κανόνες προληπτικής εποπτείας να εφαρμοστούν ομοιόμορφα σε όλα τα κράτη-μέλη ε, και σε μεγάλες επενδυτικές εταιρείες ε, και σε μεγάλα τραπεζικά ε, ιδρύματα, να πάγονται όλοι σε κοινού κανόνες εποπτείας. Τέλος, προσωπικά πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ενισχυμένη ευρωπαϊκή προσέγγιση σε σχέση με το ξέπλυμα χρήματος. Χρειάζεται ευθυγράμμιση της νομοθεσίας. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το SSM όμως ε, για να εξασφαλίσουμε συνεπή εφαρμογή σε όλα τα κράτη-μέλη. Περιμένουμε με ανυπομονησία τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. κύριος Hayes. κύριε Πρόεδρε. Και καλώς ήρθατε ξανά στην Επιτροπή μας, κυρία Νουή εκπροσωπώντα ε, τον ενίο εποπτικό μηχανισμό και σα ευχαριστώ και για τα μηνύματά σα για το ξέπλυμα χρήματο και την Τραπεζική Ένωση. Να επανέλθω στο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, ειδικά για την χώρα μου, την Ιρλανδία. Και αντιλαμβάνομαι την σημασία του να σημειωθεί πρόοδο στο θέμα για να ξεκινήσει ο δανεισμό και να βελτιωθεί η κατάσταση τη οικονομία ε, και των τραπεζών μα. Θα γνωρίζετε βεβαίως το ότι το θέμα αυτό είναι επίμαχο στην ε, Ιρλανδία, ειδικά καθώς η Alster Bank ε, πούλησε τα δάνειά της. Τρία ερωτήματα προκύπτουν. Αυτή τη στιγμή τα στεγαστικά δάνεια ε, που κατηγοριοποιούνται ως μη εξυπηρετούμενα είναι ένα θέμα Ε, που είναι χωριστά, ε, αν είναι εξυπηρετούμενα ή μη. Γιατί το εξετάζετε τόσους μήνες και δεν έχετε καταλήξει κάπου. Δεύτερον, ποια είναι η άποψή σας για το εάν η Ιρλανδική κυβέρνηση θα μπορούσε να ενισχύσει την προστασία των δανειοληπτών. Ξέρω πως είναι ζήτημα προστασίας των καταναλωτών και αφορά περισσότερο τα κράτη-μέλη, αλλά ρώτησα προσφάτως και τον πρόεδρο της ε, Κεντρικής Τράπεζας ε, και φάνηκε βεπίφορος. Τώρα, τελευταία μου ερώτηση. Έχουμε αξιολόγηση, έχουμε στρατηγική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και βεβαίως ε, τελικά υπάρχει και μια υποπτική δράση του μηχανισμού υπάρχει κάτι το ενδιάμεσο ανάμεσα στην στρατηγική και την εποπτική δράση για να υπάρχει μια διαπραγμάτευση με τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Πράγματι, το θέμα αυτό των συγκεκριμένων δανείων μας απασχολεί. Να σας πω ότι είναι ένα προϊόν ε, το οποίο διαχωρίζει το κομμάτι του δανείου εκείνου το οποίο είναι ευκολότερο να εξυπηρετηθεί από τους δανειζόμενους από ένα άλλο κομμάτι το οποίο η αποπληρωμή του εξαρτάται από τις νομικές διευθετήσεις Βεβαίως ε, το θέμα είναι περίπλοκο γιατί τα κομμάτια χαμηλής ιεραρχίας είτε εν μέρη έχουν διαγραφεί είτε έχουν διαγραφεί αλλά υπάρχει κάπου κάποιο νομικό αίτημα το οποίο ορείται άλλες φορές μπορεί να επανέλθει ε, στο κομμάτι εκείνο το οποίο είναι πιο ψηλά στην ιεραρχία των πιστωτών. Άλλες φορές υπάρχει μια έκπτωση αν εξυπηρετείται το δάνειο. Οπότε είναι περίπλοκη η κατάσταση. Συνεχίζουμε λοιπόν να εργαζόμαστε επί των θεμάτων αυτών. Καμιά φορά βεβαίως προχωράμε με διαφορετικούς ρυθμούς γιατί έχουμε 19 χώρες και αναμέναμε βεβαίως ε, τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής και τώρα που τις έχουμε λάβει μπορούμε να πούμε πως ε, εάν ε, το senior κομμάτι του δανείου αποδίδει υπό τον όρο ότι πληρούνται κάποια όροι, τότε τα δύο τμήματα του δανείου είναι τελείως ε, διαφορετικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορεί πλέον ε, να υπάρχει κάποια υποχρέωση αποπληρωμής ε, για το κομμάτι το οποίο έχει διαγραφεί μέχρι να πληρωθεί πλήρως ή να ε, χρεοκοπήσει ο δανειολήπτης ε, και αυτά ισχύουν μόνο για δάνεια Αλιανικής, ε, γιατί μόνο έτσι επιτρέπεται αυτή η προσέγγιση, ενώ για επιχειρήσεις είναι διαφορετική η προσέγγιση. Τα λέω τεχνικά, αλλά είναι και τεχνικό το ζήτημα. Εν ολίγης συμφωνούμε με τις απόψεις των Ιρλανδικών εποπτικών αρχών και μπορούμε να δεχτούμε κάποιους, ε, κάποιους λογικούς όρους ε, ότι το προϊόν βεβαίως αυτό μπορεί να τύχει αυτή τη μεταχείριση. Ναι, για το άλλο θέμα, την προστασία των καταναλωτών. Ε, αυτό επαφίεται στις εθνικές κυβερνήσεις, αν θέλουν δηλαδή να βοηθήσουν να αποπληρωθούν ε, τα δάνεια για να αποφευχθούν κάποιες αρνητικές συνέπειες και ξέρω πως υπάρχουν κάποιες χώρες που εξετάζουν κάτι τέτοιο αλλά αυτό δεν μας αφορά οι κυβερνήσεις καν ό,τι θέλουν ε, σε αυτό και δεν είναι κρατικές ενισχύσεις γιατί πρόκειται περί κοινωνικού μέτρου. Σας ευχαριστώ, Περμάνος Περές. Ευχαριστώ, κυρία Νουή, για την υπόθεση ε, της ε, Μπέλβε βλέπουμε ότι δεν είναι ικανοποιητική η κατάσταση όσον αφορά το ξέπλυμα χρήματος. Έχουμε πολλά ακόμα να κάνουμε, αλλά εγώ θέλω να επανέλθουμε στην υπόθεση ε, πτώχευσης. Ακόμα και αν δεν είναι απόλυτη η αρμοδιότητά σας, μπορεί να προτείνετε στον νομοθέτη κάποιες ε, εναλλακτικές ακριβώς ε, στο πνεύμα που έγινε και πριν από λίγους μήνες όταν αρχίσαμε να μιλάμε για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Και έπειτα ως συνεισηγήτρια για την αναθεώρηση των τραπεζικών αρχών ε, και για την υπόθεση της εποπτείας, ποια θα είναι η διάρθρωση των αρμοδιοτήτων ανάμεσα στον εποπτικό μηχανισμό και την ε, αρχή των τραπεζών, ορίστηκε αυτό σε ένα πλαίσιο που το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τοποθεσία η έδρα της ε, τραπεζικής αρχής σήμαινε ε, ότι δεν θα υπήρχε ε, πραγματική προσέγγιση ανάμεσα στην τραπεζική αρχή και τον ενιαίο υποπτικό μηχανισμό σε μια φάση όπου ο ρόλος των τραπεζικών αρχών ήταν να συμβάλλουν να σταθεροποιηθούν οι αγορές. Αυτό ήταν ο στόχο. και ποιοι είναι οι δικοί σας στόχοι σε αυτή τη μεταρρύθμιση, πώς βλέπετε να είναι αυτή η διάρθρωση να σχηματίζεται αυτή η διάρθρωση και αν αυτά τα που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, σας φαίνονται αρκετά ή επαρκή. Τελευταία μου ερώτηση. Τι γίνεται με τη σχέση των όσων εργάζονται στη ρύθμιση τη λογιστική και του ενιαίου μηχανισμού και της αρχής τραπεζών. Λέτε ότι υπάρχει μια θεσμική δομή που υπάρχει με τα φράγ. Μήπως χρειάζεται μια τάξη παρατηρητών, ένας διάλογος σε πάση περιπτώσει. Και αν ναι, πώς θα, θα πρέπει αυτό να θεσμοθετηθεί. Εγώ θα μιλήσω στα αγγλικά, αν δεν σας πειράζει ώστε να καταλάβουν περισσότεροι. Όσον αφορά την ε, πτώχευση, πολύ εκπλαγηθήκαμε που είδαμε μια κατάσταση όπου η τράπεζα είχε οριστεί ως ε, πολύ μεγάλη για να πτωχεύσει από τον ενιαίο επιπτικό μηχανισμό, αλλά τελικά ε, το νέο Συμβούλιο Εξυγίασης αποφάσισε ότι έπρεπε να γίνει αυτό και έπρεπε να ε, ε, γίνει αυτό, όμω όχι σε εθνικό επίπεδο, ούτε στη Λετωνία ούτε στο Λουξεμβούργο. Και αυτό οφείλεται στο γεγονό ότι οι Ευρωπαίοι νομοθέτες είχαν υπόψη του ότι αυτή η υπόθεση έπρεπε να ρυθμιστεί σύμφωνα με τους εθνικούς νομοθεσίες εξ, εξυγίανσης που έγινε για την Βένετο ή την Βιντζέντζα στην Ιταλία. Ε, όμως αυτό δεν είχε ρητά υποθεί. ούτε στον κανονισμό SRM, ούτε στην ΕΚΤ. E Έπρεπε δηλαδή το κράτος να έχει καταλάβει ότι αυτό εννοούσε αν και εάν δεν το αναγνωρίσουν οι... τα κράτη δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ε, στο έπακρο τους κανονισμούς αυτούς. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αυτό πάει στους εθνικούς ε, δικαστές που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά τις εθνικές νομοθεσίες και ποια είναι τα κριτήρια τα οποία ε, πυροδοτούν την εξυγίανση. Και δεν μπορούν να πιστούν από κάτι το οποίο υπονοείται από μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει ρητά να γραφτεί στην ευρωπαϊκή νομοθεσία ότι μία τράπεζα πρέπει να εξηγενθεί σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. Οι δικοί μου νομική σύμβουλοι μου λένε ότι το άρθρο 32 ε, της ε, οδηγίας DRD είναι το καλύτερο. Και ότι Αυτά θα πρέπει να συνοδευτούν από εθνικές ενέργειες ώστε να προσθεθούν τα κριτήρια εξηγήσεω για τις τράπεζες. Μόνο για τις Τράπεζε, είναι περιορισμένος πληθυσμό δηλαδή, δηλαδή η δήλωση του ενιαίου επιπτικού μηχανισμού και η επιβεβαίωση από τον SRM. ο ρόλος ανάμεσα στην αρχή των τραπεζών και στον ενιαίο εποπτικό μηχανισμό. Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών θα μπορούσε να είναι ο Ευρωπαίος επόπτης, όμως δεν εκρίθη αυτό αρκετό. Υπάρχει ο Ευρωπαϊκός Εποπτικός Μηχανισμός που είναι υπεύθυνο και αρμόδιος για την εποπτεία σε ολόκληρη την Ευρωζώνη. Όταν μιλάμε για, την Ευρωπαϊκή, για το Εποπτικό Συμβούλιο τη αρχή των Τραπεζών είναι πολύ σημαντικό ο ρόλος του γιατί ειδικά για εμά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε 19 εθνικά πλαίσια είναι πολύ καλό λοιπόν που έχουμε το Εποπτικό Συμβούλιο ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνοχή σε όλα αυτά αλλά προφανώς το όριο στην εποπτεία είναι οι δοκιμέ αντοχής, τα stress test που γίνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο. Για το ενιαίο Συμβούλιο Εξυγένσης εμείς ε, στηρίζουμε την πρόταση που γίνεται. Θεωρούμε πως έχει νόημα να στηρίξουμε το προσωπικό ώστε να πάει στην έκτε κοντά, έτσι θα μπορούν να συνεργάζονται καλύτερα και ε, για τη λογιστική έλεγχο, ναι, συνεργαζόμαστε και, ε, συν, με την ΦΡΑΓ. Είναι πολύ θετική συνεργασία, αλλά κάθε είδου συνεργασία και συντονισμός είναι θετικός. Για να είμαι ειλικρινής, Έχουμε καλές συζητήσεις με τους ε, ε, ελεγκτές ε, με τις τράπεζες τις οποίες εποπτεύουμε μία-δύο φορές το χρόνο, ανάλογα με την κατάσταση. Και αυτό είναι επίσης πηγή ανταλλαγών θετικών. για να μπορούμε να εξηγήσουμε τις απόψεις μας. Είμαστε μέρος του διαλόγου λοιπόν και το Εποπτικό Συμβούλιο είναι μέρος αυτού του διαλόγου. Λούντς. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κυρία Νουή που είστε εδώ σήμερα. Αναφέρατε στην εισήγησή σας ότι περισσότερη ρύθμιση για τις τραπεζικές ρυθμίσεις ε, χρειάζονται. Πολύ ενδιαφέρον αυτό, ειδικά εφόσον ε, δώσατε συγκεκριμένη απάντηση στην ερώτηση της συναδέλφου Μπερές που μάλιστα κάνατε μία ε, συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για την BRD. Πάντοτε είναι ενδιαφέρον να ακούμε τι προτάσει αυτέ από εμπειρογνώμονε, ιδιαίτερα όσον αφορά την μείωση του κινδύνου. Πριν από δύο εβδομάδε είχαμε την πρόταση ε, τη ε, Κομισιόν για τροποποιητικό κανονισμό του CRR, του Κανονισμού Κεφαλαιακών Απαιτήσεων, για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πρέπει δηλαδή κάπως να χειριστούμε το τεράστιο στόκ των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχει μέχρι σήμερα. Ε, εγώ ε, θέλω να σας ρωτήσω, είστε ικανοποιημένοι με αυτή την πρόταση, αυτό περιμένατε και αν είχατε δική σας επιλογή, εσείς την επιλογή, τι θα κάνατε ακριβώς, πώς θα το συνεχίζετε αυτό. Και νομίζετε ότι αρκεί αυτή η συμβολή της Κομισιόν για τη μείωση του κινδύνου, γιατί για να είμαστε ειλικρινείς είχαμε διάφορες προτάσεις. Αλλά Διαρωτώ με χρειάζονται περισσότερες. Αν κοιτάξουμε την, ε, τον πρώτο πυλώνα, θα δείτε ότι ισχύει μόνο για τα νέα δάνεια και όχι ε, για τα παλιά δάνεια. Αν με τη νέα οδηγία, έχουμε την ανάκτηση ε, των δανείων στη, όχι στη, μόνο στη δευτερογενή αγορά Βλέπουμε λοιπόν ότι κάποιες προτάσεις είναι επιθελοντικής βάσης. Η ερώτησή μου είναι αν κάνουμε αρκετά και αν αυτό που κάνουμε τα κάνουμε σωστά. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί η Βασιλεία 3, πρέπει να εφαρμοστεί βεβαίω για τη θεμελιώδη αναθεώρηση του Trading Book, το οποίο εκκρεμεί εδώ και καιρό. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να μεταγραφεί σε ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αναφέρατε την αλλαγή στην ε, BRD για να εξασφαλίσουμε την εξυγίανση τραπεζών όταν δεν... Ε, ε, μάλλον την εκαθάριση τραπεζών σε περίπτωση που δεν μπορούν να εξυγιανθούν. Ε, γιατί εκεί έχουμε ε, θέμα σταθερότητας, αλλά να έχουμε μεγαλύτερες τράπεζες που διατηρούνται σε αυτή την κατάσταση τη μετέωρη, που ε, πτωχεύουν, αλλά είναι πολύ μεγάλη για να πτωχεύσουν, αλλά δεν καθαρίζονται και δεν εξηγένονται. Εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να δούμε και τη διαδικασία αυτό Εμεί Εμείς θέλουμε, αυτή η διαδικασία δεν είναι τόσο ικανοποιητική, θα πρέπει να υπάρχει δικαστική ε, διαδικασία. Αυτή είναι η πιο σημαντική. Εγώ θα έλεγα ότι ο πρόεδρος ε, του ενιαίου συμβουλίου θα έπρεπε να είναι μέλος ε, του ενιαίου μηχανισμού εξυγίανσης, γιατί υπάρχουν διάφοροι ιδρύματα τα οποία δεν πιστεύουν όταν τους λέμε ότι συνεργαζόμαστε πλήρως με το ενίο Συμβούλιο Εξυγίασης. Απόλυτη απόδειξη θα ήταν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι με τα μέλη μας. Ήταν δύσκολο να πούν τότε ότι δεν υπάρχει ελεύθερη ροή πληροφοριών. Και επίση θεωρώ ότι είναι κάτι εύκολο να γίνει. Όσον αφορά την μείωση του κινδύνου, Πολλά έχουν γίνει ήδη. Συνεχίζεται η προσπάθεια για τα κόκκινα δάνεια. Και κατά τη γνώμη μου, η αλληλεγγύη για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης θα πρέπει να κινηθεί παράλληλα με τη μείωση κινδύνου, ώστε να μοχλεύουν αλλήλους. Αυτό που βλέπω όμως ότι είναι σημαντικό, εξίσου σημαντικό σχεδόν με το μείωση του κινδύνου, είναι η ο σημερινός κατακαιρματισμός του νομικού πλαισίου εντός της Ευρώπης. Χρειάζεται περισσότερη εναρμονισμένη νομοθεσία, λιγότερες εθνικές επιλογές, περισσότεροι κανονισμοί από ό,τι οδηγίες υπόθεση που αφορά την καθάριση, την πτώχευση, σημαίνει, είναι επίση θέμα νομικής, νομικού κατακαιρματισμού. Αυτό είναι πραγματικό εμπόδιο στο να ωφεληθούμε από την Τραπεζική Ένωση. Ο, λείπει και ο πυλώνας 3, ναι, αλλά και ο κατακαιρματισμός της νομοθεσίας είναι επίσης πρόβλημα. Thank you, Ramon Grazie, Presidente. Ε, ε, Γεια σας κύριε Νουή, καλώς ορίσατε και πάλι δύο ερωτήσεις έχω. Για τη ΜΥΦΗ 3, ε, κάποια κράτη-μέλη ανησυχούν για τη συγκέντρωση στην αγορά για τις μεγάλες τράπεζες και τους μεγάλους διαχειριστές στοιχείων ενεργητικού, διότι είναι αυξανόμενο το κόστος για τη διαφάνεια και για την λογοδοσία οι μικρομεσαίοι μάνατζες και οι μικρομεσαίες τράπεζες πώς μπορούν να αποτρέψουν κάτι τέτοιο. Και δεύτερον, για τα κόκκινα δάνεια. Ε, Μπορεί κάποια κράτη-μέλη, το αντιλαμβάνομαι, να μην θέλουν να μειώσουν το ε, περιθώριο για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Αλλά έχουμε για τα αλλά και το κανονισμό για τη δευτερογενή αγορά και ε, ξέρουμε και τι γίνεται με το blueprint. Πολύ ωραία όλα αυτά. Όμω, τη ρίζα του κακού δεν την αντιμετωπίζουμε στα κράτη-μέλη. Δηλαδή, ε, τις οδηγίες για τις καθυστερούμενε πληρωμέ δεν τι εφαρμόζουν σωστά. Ε, ε, αυξάνονται τα επιτόκια Αν δεν πληρώνουν ε, φερέγγες ε, δεν πληρώνονται εγκαίρως ε, φερέγγες σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τις μεγάλες τις επιχειρήσεις, τότε θα έχουμε άλλο ένα κύμα, άλλο ένα τσουνάμι κόκκινο. Τι πιστεύετε εσείς. Κοιτάξτε η συγκέντρωση των αγορών για τις τράπεζες και για τους asset managers. Ε, είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, ε, διότι στην πρώτη περίπτωση εξαρτάται από τη χώρα. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ε, εμφανίστηκαν κάποιες λόγω της κρίσης. Είναι κρίμα, αλλά αυτό συνέβη. Όμως, Εάν θεωρήσουμε ως ενιαία δικαιοδοσία το SSM και λένε και περισσότερο αυτό θα έπρεπε να κάνουμε, κυρίως θα ολοκληρωθεί η Τραπεζική Ένωση με τον τρίτο πυλώνα, τότε Αυτό το επίπεδο συγκέντρωσής δεν θα είναι τόσο υψηλό, διότι θα αυξηθούν ε, οι μικρές και μεσαίε ε, τράπεζες. Ε, θα υπάρχει μεγαλύτερη πυκλομορφία, Θα έχουμε και τράπεζες που δεν είναι στο χρηματιστήριο, θα έχουμε συνεταιριστικέ τράπεζες και μικρές, μικρές τράπεζες και το καθεξής. Λοιπόν, αυτή η πυκλομορφία υπάρχει και αποτυπώνεται και στη, στους κανονισμούς. Για τους asset managers είναι διαφορετική κατάσταση. Μας ε, βοηθάει το μέγεθος για να μπορούμε να τιμολογήσουμε σωστά τις ε, υπηρεσίες. Για να διατηρήσουμε και την ανταγωνιστικότητα αυτών των managers, αυτών των διαχειριστικών εταιριών. Δεν νομίζω ότι θα προκύψει αυτό το κύμα που είπατε συγκέντρωσης. Είναι πολύ καλό λοιπόν για τα NPL, για τα κόκκινα δάνεια που έχουμε τόσο πολλά εργαλεία για να τα αντιμετωπίσουμε ούτως ώστε να μπορούμε να αποφύγουμε φαινόμενα όπως αυτό που παρατήσαμε, δηλαδή να σχεδιάσετε ένα νέο προϊόν, δηλαδή παίρνετε αυτό που μπορείτε να σώσετε από το κόκκινο δάνειο και μετά με την ε, οριμότητα του δανείου αποφασίζετε να δημιουργήσετε ένα νέο προϊόν. Πολλές λύσεις υπάρχουν, εξαρτώνται όλα από τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, αν ε, είναι για επιχειρήσεις ή για ε, ιδιώτες, αν ε, έχουν την έδρα τους ή δεν την έχουν στο κράτος μέλος και το καθεξής. Και με το παράρτημα αυτό κάνουμε, αποφεύγουμε τη συσσόρευση νέων ε, κόκκινων δανείων και σίγουρα θα τροποποιήσουν τα κριτήρια τους οι τράπεζες για την ε, ε, πίστη, ούτως ώστε να είναι ασφαλή τα δάνεια και μην ξεχνάμε ότι είναι οικονομικέ οικονομικές ε, προϋποθέσεις ε, όταν ε, συνάπτονται αυτά τα δάνεια. Όχι όταν όλοι θέλουν να αποφύγουν το δάνειο και τον κίνδυνο που συνεπάγεται επειδή ούτω ή άλλως υπάρχει κρίση. Αυτό που με ρωτήσατε για τις φερέγγιες ε, μικρομεσαίες. Ε, φυσικά είναι κλειδί. Πρέπει οι πελάτες να τις πληρώνουν ε, και ε, δεν αποκλείει και το δημόσιο από αυτό. Ε, πρόθεσμα πρέπει να πληρώνονται. Και πρέπει να βρουν τραπεζικά προϊόντα σε λογικές τιμές για να μην δημιουργήσουν περαιτέρω εκθέσεις ε, μη εξυπηρετούμενες. Γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο για τις ε, τράπεζες, αλλά και για τις εταιρείε, ε, για τις επιχειρήσεις που δανείζονται. Γιατί άμα δεν τα αποπληρώνουν, δεν θα πάρουν καινούργια δάνεια. Οπότε, ναι, όντως θα πρέπει να ε, επικρατήσει αυτή η κουλτούρα και να υπάρχουν τα κατάλληλα τραπεζικά εργαλεία, πέρα δηλαδή από το κανονιστικό πλαίσιο για τα κόκκινα δάνεια, να υπάρχει μια διαδικασία ούτω ώστε τα μη εξυπηρετούμενα να γίνονται εξυπηρετούμενα τουλάχιστον ε, στην αρχή, ούτως ώστε για το μέλλον να έχουμε καλύτερα δάνεια. Ευχαριστούμε, Σβέν Γκίγκολ. Κυρία Νοή τις τελευταίες εβδομάδες ε, και μήνες ε, μια σειρά τραπεζικών εγκλημάτων στην Τραπεζική Ένωση. Στην Μάλτα είδαμε τον διαφήνοντα συμβουλό της Τράπεζας Πιλάτους που έχασε το δικαίωμα να ασκήσει τα δικαιώματά του στις μετοχές της τράπεζας μόνο κατόπιν αμερικανικών πιέσεων. Είδαμε την θηγατρική της Danske Bank στην Εστονία. Έχουμε και άλλα προβλήματα εκεί πέρα εξεπλήματος χρήματος και στη Λετωνία η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα υπό την άμεση υποπτία σας περιγράφεται από το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών ως εξής. Οι περισσότεροι πελάτες της εταιρείας είναι εταιρείες γραμματοκιβώτια με έδρα εκτός Λετωνίας. Και συνεχίζω. Η διοίκηση της τράπεζας ε, προσπαθεί να εμποδίσει την εφαρμογή των κανόνων της ε, χώρας ε, καθ' όλη τη διάρκεια του 2017. Τα στελέχη της τράπεζας χρησιμοποίησαν δωροδοκίες για να επηρεάσουν στελέχη του κράτους όταν διερευνούσαν ε, τις δραστηριότητες της τράπεζας και τα λοιπά και δεν ασκεί σωστά την πολιτική know your customer και σύμφωνα με την ίδια την αξιολόγηση της τράπεζας το μεγαλύτερο ποσοστό των πελατών της είναι υψηλού κινδύνου εταιρείε γραμματοκιβώτια που είναι εγγεγραμμένες σε μυστικές ε, ε, σε άλλες χώρες οι οποίες ε, δεν γνωρίζουν ποιες είναι. Κυρία Νουή, μήπως ε, να φέρουμε τις ΗΠΑ να ασκούν εποπτεία στην Τραπεζική μας Ένωση. Ζητάτε περαιτέρω ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα στην εκθεσή σας, αλλά μπορεί, και συμφωνούμε, μπορείτε όμως να δεσμευτείτε ότι χρησιμοποιήσετε τα μέσα που έχετε ήδη στην διάθεσή σας για να καταπολεμήσετε το οικονομικό έγκλημα στην Τραπεζική Ένωση και ποια νέα μέσα θα και πόρους θα αφιερώσετε για να συνεισφέρετε στην καταπολέμηση του ξεπλήματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Όπως γνωρίζετε και εσείς ε, και αρκετοί, ο κανονισμός του ενιαίου υποπτικού μηχανισμού περιέχει την ε, απόφαση συνειδητή του Συμβουλίου να μην δώσει αυτές τις αρμοδιότητες περί ξεπλήματος χρήματος ε, κλπ. στην Κεντρική Τραπεζά. Υπάρχουν όμως κάποιες ε, στιγμές ε, όπου πλησιάζουμε εκεί ή συμπίπτουν οι ενέργειές μας, όπως παραδείγματο χάρη όσον αφορά τις τραπεζικές αδείες. Τούτου λεχθέντος η παραβίαση των νόμων περί ξεπλήματος χρήματος δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Μόνο αν έχουν αποδειχθεί τέτοιες περιπτώσεις από τις αρμόδιες αρχές, μπορεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να θεωρήσει ότι αυτά είναι δεδομένα και να χρησιμοποιήσει τις παραβιάσεις αυτές είτε για αφαίρεση της αδείας είτε για δράσεις ε, του πυλώνα 2. Όμως ε, τέτοια μέτρα έχουν ε, περιορισμένο μέγεθος γιατί τα μέσα αυτά δεν είναι τα καταλληλότερα για την παρακολούθηση ξεπλήματος ε, χρήματος ή ακόμα και η έλλειψη εσωτερικών ελέγχων που επιτρέπει σε αυτούς που κάνουν αυτή τη δουλειά να χρησιμοποιούν τις τράπεζες για ξεπλήμα χρήματος. Συμφωνώ ε, Πράγματι είναι άσχημη εικόνα να βασιζόμαστε στη ΣΥΠΑ και πρέπει να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Ευχαρίστω, εγώ δεσμεύω να κάνω ό,τι μπορώ, αλλά όπως σας είπα αυτά τα κάναμε ήδη, δεν ήταν επαρκή και αμφιβάλλω εάν θα είναι επαρκή στο προσεχές μέλλον. ευχαριστώ το ότι θα υπάρξει μια πέμπτη οδηγία για το ξέπλυμα χρήματος που τουλάχιστον θα ξεκαθαρίσει το ότι μπορούν να υπάρχουν ανταλλαγές πληροφοριών από τις εθνικές αρχές που είναι αρμόδιες για το ξέπλυμα χρήματος ε, με εμάς. Κάτι το οποίο δεν είναι ερητό αυτή τη στιγμή και βασιζόμαστε μόνο στην καλή θέληση των εθνικών αυτών αρχών. Προφανώς ε, και εμείς ε, όταν βρίσκουμε σε επιτόπιες επιθεωρήσεις για προληπτικούς σκοπούς, όταν βρίσκουμε κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι ε, ποινική υπόθεση, τα στέλνουμε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος μετά θα αποφασίσει αν υπάρχει κάτι προς διοξινή ή όχι. Αλλά είμαστε σε καλύτερη θέση με την εφαρμογή της πέμπτης οδηγίας ξεπλήματος χρήματος, αλλά προσωπικά ε, θεωρώ ότι αυτό δεν αρκεί Χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό θεσμικό όργανο το οποίο θα εφαρμόζει με τρόπο συνεπή την νομοθεσία αυτή στην Ευρωζώνη. Γιατί καμιά φορά έλεγα ότι οι μικρές χώρες ε, δεν έχουν αρκετό προσωπικό ή πείρα όταν αντιμετωπίζουν ε, κάποιες αρκετά σοβαρές ε, πιθανότητες ε, ξεπλήματος ε, χρήματος. Οπότε, ναι, πρέπει να αλλάξει η κατάσταση που δεν μπορούμε πια να είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Σα Σας ευχαριστώ. Μάρκο Βάλλη. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αν θέλετε να βάλετε τα ακουστικά σας, γιατί θα μιλήσω στα Ιταλικά. Σας ευχαριστώ. Τι, ποια είναι η άποψή σας για τη δημοσίευση προς, ε, προσαρτημάτων που, έχουν, που έχει ε, οδηγήσει σε πολλές συζητήσεις, έντονες συζητήσεις. Μισό λεπτό, μισό λεπτό περιμένετε παρακαλώ. Εντάξει τώρα. Έλεγα λοιπόν Ποια είναι η αποψή σας για τη δημοσίευση του προσαρτήματος που δημιούργησε ε, διάφορες συγκρούσεις και άναψε τη συζήτηση για το κομμάτι αυτό που συνδέεται με τα κόκκινα δάνεια. Λειτουργεί, με ακούτε, γιατί είμαστε σε μια κατάσταση όπου εφαρμόζεται μια διαδικασία που οδηγεί τις τράπεζες να ζητούν πολύ περισσότερες εγγυήσεις για να μπορέσουν να δώσουν ε, δάνεια στη πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στις οικογένειες, στους ανθρώπους που συμβάλλουν ε, περισσότερο στην ανάπτυξη και στην οικονομία και έτσι δεν δημιουργείται κίνητρο αλλά ε, συρρήκνωση. Στη στιγμή που η ανάπτυξη στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη και ιδιαίτερα στι νότιε χώρες που έχουν ε, τραπεζικά μοντέλα πολύ εκτεθειμένα στο σύστημα της πίστοση θα οδηγήσει σε συρρήκνωση και μάλιστα θα οδηγήσει τι τράπεζες σε περίπτωση μελλοντικών κρίσεων να πρέπει να ε, καθαρίσουν αντί να διαχειρίζονται τις ε, πιστώσεις φθαίρετα. Δηλαδή τα κερδοσκοπικά ταμεία τα οποία αυτή τη στιγμή ε, καθοδηγούν την αγορά, αυτά κερδίζουν περισσότερο. Και δεν είναι εύκολο να γίνει κάτι τέτοιο για τα κόκκινα δάνεια. Πώς μπορείτε να δημοσιεύετε ένα τέτοιο πράγμα χωρίς πρώτα να έχετε δημοσιεύσει μια αξιολόγηση αντικτύπου για την ιδέα σας αυτή, ποσοτικά και ποιοτικά. Όταν δηλαδή κάνετε τέτοιου είδους προτάσεις, κάνετε αξιολογήσεις ή το εφαρμόζετε έτσι απλά και μόνο επειδή έχετε την πρόθεση να εξαλείψετε το πρόβλημα των ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων χωρίς να καταλάβετε ποια είναι η συγκεκριμένη κατάσταση, χωρίς να καταλάβετε ότι θα δημιουργήσετε πρόβλημα στο σύστημα πίστοσης που θα έπρεπε να προσεχθεί ιδιαίτερα. Ενώ η χρηματοπιστωτική αγορά, η κεφαλαία αγορά, ας πούμε, οι τίτλοι τρίτου επίπεδου ε, έκθεσης δεν το έχετε ακόμα, δεν σας έχει απασχολήσει. Θέλω να ξέρω λοιπόν αν κάνατε αξιολογήσεις αντικτύπου και αν θέλετε να δημοσιεύσετε αυτά σε σχέση με το ε, ε, προσάρτημα. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Το να είναι αποδοτικά τα δάνεια και να αποπληρώνονται δεν σημαίνει απαραίτητο περισσότερες εγγύησεις. Από τη στιγμή που η ανάκτηση των collateral είναι αργή σε, με συγκεκριμένα νομικά πλαίσια και συγκεκριμένες χώρες. Κατά τη γνώμη μου, το θέμα είναι να είναι καλύτερη, καλύτερα τα κριτήρια εγγύησης ε, ε, για την ε, χορήγηση δανείων. Καλύτερη εποπτεία της κατάστασης της δανειοδότησης, γιατί όταν κανείς παρέμβει νωρίς, δεν είναι τόσο περίπλοκο το να αναδιαρθρώσει το δάνειο ώστε αυτό να συνεχίσει να αποδίδει εφόσον κάτι τέτοιο χρειάζεται σε σχέση με τη συρρήκνωση της παροχής πιστώσεων εδώ και αρκετά χρόνια τώρα δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί στο μέλλον να επανέλθει, αλλά για την ώρα έχουμε κατάσταση και στην Ιταλία και αλλού που δεν ε, δείχνει συρρήκνωση και γι' αυτό ακριβώς ε, είναι η κατάλληλη στιγμή να εξασφαλίσουμε ότι ε, οι τράπεζες θα ασχοληθούν με, το με τα αποθέματά τους. Για να σταθεί η οικονομία χρειάζεται να έχουμε σταθερές και ισχυρές τράπεζες, όχι να αγωνίζονται να επιβιώσουν. Επίσης, η ισόρρευση νέων μη εξυπηρετούμενων δανειών θα πρέπει να σταματήσει. Και δεν μπορούμε να πούμε ήδη ότι η παροχή μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει σταματήσει στις χώρες που ήδη είναι επιβαρημένες. Είπατε ότι προσέχουμε υπερβολικά αυτό το θέμα. Όταν ξεκινήσαμε με τον ε, εποπτικό μηχανισμό είχαμε ένα τρισεκατομμύριο μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις χώρες ε, αυτές. τώρα έχουμε φτάσει στα 700 δις, που πάλι είναι πολύ μεγάλο νούμερο. Οπότε κάτι πρέπει να γίνει. Δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν, δεν γίνεται να μην ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Αυτό που κάναμε μέχρι τώρα με το προστατικό στις, στις οδηγίες ε, ε, ακόμα αφορά τα πρώτα στάδια. Θέλουμε να ενεργήσουμε πριν δηλαδή το πρόβλημα γίνει μεγαλύτερο. Δεν χρειαζόταν ε, νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Υπήρχαν κάποιοι που υπολόγισαν τι θα σήμαινε, αλλά όχι πολύ ε, επισταμένος. Πού είναι η αξιολόγηση αυτή ε, αντικτύπου στην πραγματική οικονομία. Αυτό θα έπρεπε να γίνει αν χρησιμοποιούσαμε το, προσάρτημα για για το απόθεμα. Εκεί μπορούμε να κάνουμε ε, ε, αξιολόγηση αντικτύπου, γιατί ξέρουμε ποιο είναι το απόθεμα. Αλλά για τα ε, νέα κόκκινα δάνεια δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, τα οποία μπορούμε δηλαδή να τα μετατρέψουμε σε αποδοτικά. Κάτι τέτοιο δεν είναι σκόπιμο, ούτε καν εφικτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Ναι, θα ήθελα πολύ να οριστούν αυτά στις οικονομίες όπου είναι επιβαρημένες με μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Όταν αυτή η υπόθεση τελειώσει θα είναι πολύ καλύτερη κατάσταση. Σας ευχαριστώ. Ε, αυτό το οποίο λέτε ότι δεν έχουμε μείωση της παροχής ε, πριν τεθούν τα μέτρα ενισχύ, ε, θα έπρεπε να το πείτε αντίστροφα. Γιατί δεν λέει τίποτα για το ότι τα νέα μέτρα θα επηρεάσουν την τραπεζική πιστή ακόμα δεν έχουν τεθεί ενισχύ. Τέλος δεν το αντιλαμβάνουμε αυτό το οποίο λέτε. Ο κύριος Τζάνι. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσείς ε, Αναφέρατε νούμερα για να αιτιολογήσετε αυτόν τον ζήλο από πλευράς του μηχανισμού επεπτείας για τον ε, κίνδυνο της πίστοσης ανάλυσης και διατάξεις που ε, έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια. Εγώ, ωστόσο, βλέποντα τα νούμερα των ισολογισμών των τραπεζών υπό την άμεση υποπτία τη ε, ΕΚΤ, βλέπω να εξακολουθεί να υπάρχει μια μεγάλη ασυμμετρία ε, στην αντιμετώπιση του κινδύνου πίστοσης και, του, και της αγοράς. Βλέπουμε για τίτλους επίπεδου 2, επίπεδου 3 που υπάρχουν στις τράπεζες, ειδικά στα μεγάλα ιδρύματα της Βόρειας Ευρώπης. Εσείς αναφέρατε το 1-3 των ε, κόκκινων δανείων στις τράπεζες όταν ξεκινήσατε τη δραστηριότητά σας. Εγώ σας παραθέτω ότι είναι πέντε-τρεις ε, η αξία αυτών των τίτλων που έχουν τεράστιο βάρος ε, ως ε, στοιχεία ενεργητικού. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο ενιαίος ευρωτικός μηχανισμός εξακολουθεί να υποτιμά αυτό το κίνδυνο και η τάση είναι ότι δημιουργείται μια συμμετρία που κάνει διακρίσεις ανάμεσα στα εθνικά συστήματα και δίνει, και δίνει πιο βολική τη λύση ε, την προφύλαξη από τους κινδύνους σε σχέση με την πραγματική χορήγηση δανείων στην πραγματική ε, οικονομία. Και έτσι ε, αφήνει, μόν, αφήνει απείρευτο έναν από τους πιο σημαντικούς παράγοντες, ε, λόγους μάλλον για την κρίση. η δραστηριότητα του επόπτη θα επικεντρωθεί στο κίνδυνο στην αγορά και θα ληφθούν ε, συγκεκριμένα μέτρα ώστε να εξοδετερωθεί αυτός ο κίνδυνος που δεδομένων των νούμερων των ισολογισμών μπορεί όντως να θέσει υπό, ε, υπό, σε πρόβλημα, να δημιουργήσει προβλήματα μάλλον στο ευρωπαϊκό σύστημα. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Δεν ε, συμφωνώ με την αξιολόγηση ότι δεν κάνουμε εξίσου καλές ελέγχους για την αξιολόγηση των μοντέλων των τραπεζών για το επίπεδο 3 και επίπεδο 2 μάλιστα, που είναι εξίσου σημαντικό. Ερευνούμε τις πτυχές του ρίσκου της αγοράς σε τακτική βάση και βεβαίως αυτά αναφέρονται στην αξιολόγηση κινδύνου της ε, αγοράς. Έχουμε κάποιες ε, επιτόπιες επίσης επιθεωρήσεις. Έχουμε κάποια οριζόντια μέτρα σύγκρισης με βάση τα οποία κάνουμε την ανάλυση με τρόπο συνεπή και εγώ θα έλεγα πως ε, η λειτουργία της αγοράς ε, χρησιμοποιούνται δύο φορές ως ε, κριτήρια για τις παγκόσμιους εκείνους κανόνες που αφορούν το επιπλέον, τις επιπλέον κεφαλαϊκές απαιτήσει. και αυτό σημαίνει ότι απαιτείται πλέον κεφάλαιο για την πολυπλοκότητα και επιπλέον κεφάλαιο λόγω του στοιχείου της διάσωσης γιατί αν δεν υπάρχει μια αγορά για κάτι τέτοιο τότε είναι πιο εύκολη η διάσωση του των δεν θα έλεγα ότι δεν στηρίζουν την οικονομία η αγορές των τραπεζών ε, για λογαριασμό τους έχουν μειωθεί πάρα πολύ λόγω της ε, κρίσης. Μεγάλο κομμάτι ε, των λειτουργιών είναι απλά παράγωγα που χρειάζονται οι τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις για να συμμετέχουν στην οικονομία. Ίσως έχετε επίσης παρατηρήσει ότι ζήτησα το Κοινοβούλιο τους νομοθέτες να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν αυτό το οποίο λέμε μια ουσιαστική εξέταση του trading book, δηλαδή να δούμε ακριβώ ποιες είναι αυτές οι λειτουργίες της αγοράς ε, που απαιτούν επαρκές κεφάλαιο πριν ή κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης. Ελπίζω να συμβεί αυτό λοιπόν, αν θέλετε να συνεισφέρετε σε αυτήν την αύξηση κεφαλαιακών απαιτήσεων. Νομίζω ότι κατά την άποψή μου έτσι πρέπει να προχωρήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο πρέπει. Αντέλος. Ευχαριστώ κύριος Σκίτσος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω την εντύπωση ότι τα πάμε πολύ καλά όσον αφορά την μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι μεταξύ άλλων κάνετε καλή δουλειά. Θεωρείτε ότι φτάνουμε σε ένα χαμηλό επίπεδο μη εξυπηρετούμενων δανείων που θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της διαδικασίας τραπεζικής ένωσης ή πρέπει να συνδυάσουμε ένα χαμηλότερο μεσόωρο με συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως την Ελλάδα ή την Κύπρο από τις μικρότερες χώρες και την Ιταλία από τις μεγαλύτερες. Και άλλη μία ερώτηση για την Ελλάδα. Φαίνεται ότι η επικρατούσα άποψη στην Ελλάδα είναι ότι ο τραπεζικός τομέας πηγαίνει καλύτερα, αλλά ταυτόχρονα πολλοί αναλυτές και πολιτικοί και οικονομολόγοι θεωρούν ότι αυτή η βελτίωση της κατάστασης ε, πρέπει να επιταχυνθεί έτσι ώστε ο τραπεζικός τομέας θα βοηθήσει περισσότερο την χρηματοδότηση της ανάπτυξης του ιδιωτικού τομέα. Βλέπετε λοιπόν κάποιο σενάριο με επιπλέον μέτρα για να επιταχυνθούν οι θετικές εξελίξεις στην Ελλάδα ή θα επιμείνετε σε μια σταδιακή προσέγγιση. Ευχαριστώ. Θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε ένα ενιαίο καθεστώς για μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις ε, διάφορες χώρες της ε, Ευρωζώνης. Δεν θεωρώ ότι μπορούμε να έχουμε ε, διαφορετικά μέτρα όταν δεν έχουμε διαφορετική νομοθεσία για τις ελληνικές τράπεζες και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Πράγματι έχει σημειωθεί αρκετή πρόοδος, τώρα αν είναι αρκετά γρήγορη. Όχι ακόμα. θα έλεγα πως πρέπει να επιταχυνθεί ο ρυθμός και για όλες τις τράπεζες η στιγμή της αλήθειας θα είναι τα stress test της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής. Εκεί θα δούμε εάν οι τράπεζες αυτές και άλλες μπορούν να αντέξουν σε κραδασμούς ε, ε, που περιέχονται στα χειρότερα σενάρια, διατηρώντας ταυτόχρονα τις ε, κεφαλαίκες τους απαιτήσει. Αυτή θα είναι νομίζω η στιγμή της αλήθειας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λουίτζι Μόργανο. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε κυρία Νουή. Με συγχωρείτε αν είμαι πολύ ευθύς στην παρέμβασή μου, τι θέλω να πω. Κανονικά τα μέτρα τα οποία ε, εσείς ε, θεσπίζετε μέσα στο ρόλο σας ε, του επόπτη θα έπρεπε να συνδυάζονται με τα μέτρα που υιοθετούνται από τον νομοθέτη. Έχω την εντύπωση και μάλιστα το Κοινοβούλιο το τόνισε ότι ο θεσμός τον οποίο εσείς εκπροσωπείτε έχει μία τάση να μας βάζει ενώπιον τετελεσμένων. Πριν από την διαβούλευση για το προσάρτημα που βάλατε στο κόκκινα δάνεια ε, και με την τελική εκδοχή του παραρτήματος που δημοσιεύσατε το περασμένη εβδομάδα δεν ε, μας διαβουλευθήκατε. Αυτό το παραρτήμα έχει διάφορες σημαντικές, περιέχει διάφορες σημαντικές διαφορές σε σχέση με την πρόταση της Κομισιόν και ας μου το επιτρέψετε μπορεί να παρουσιάζει προφίλ που δεν είναι τα βέλτιστα αναδρομικά όσον αφορά την εκτίμηση των τραπεζών τραπεζών. ρωτώ λοιπόν, Πώς λοιπόν θα έπρεπε ο χρονισμός αλλά και η ουσία του παρατήματος θα επιβαρύνουν ε, την, τον τρόπο που λειτουργούν ε, οι νομοθέτε, δηλαδή το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πέρα από την ενδεικτική φύση των μέτρων που περιέχει το ίδιο το παράρτημα και έπειτα Μέχρι στιγμής ήταν αργή η διαδικασία. Τι αξιολόγηση κάνατε στην σε σχέση με την πιθανή ε, προκυκλικότητα των μέτρων που μπορεί να οδηγήσουν σε συρρήκνωση των πιστώσεων και άρα σε λιγότερη ε, ρευστότητα για τις επιχειρήσεις και άρα τον κίνδυνο να περιοριστεί το τραπεζικό δανεισμός ε, κυρίως για εκείνους που όχι πάντοτε που δεν καλύπτονται πάντοτε αρκετά καλά. Ευχαριστώ και εγώ σας ευχαριστώ. Η διαβούλευση που αναφέρατε ανάμεσα στην Επιτροπή και το παράρτημα του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού ναι, ανακοινώθηκε την ημέρα μετά της Κομισιόν. Ε, υπήρξε απόλυτο συντονισμός ε, και κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, δεν υπάρχει καμιά αντίφαση ανάμεσα στα δύο μέσα, τα οποία είναι συμπληρωματικά, παραπληρωματικά μάλλον. Εμεί καλωσορίζουμε το backstop της Επιτροπής για τα νέα δάνεια, πύλωνα 1, που θα είναι υποχρεωτικό για όλες τις τράπεζες, αλλά είναι φυσιολογικό. Ο δεύτερος πυλώνας, που είναι για κινδύνους πάνω από το μέσο κίνδυνο, που περιλαμβάνεται στο πυλώνα 1, είναι διαφορετικά και ξεκινούν σε διαφορετικό επίπεδο χρησιμοποιούνται στον εποπτικό διάλογο για συγκεκριμένες περιστάσεις όπου ο κίνδυνος είναι ψηλότερος από τον μέσο κίνδυνο που καλύπτεται από τον πρώτο πυλώνα. Αυτό είναι ο κανονικός ορισμός του δεύτερου πυλώνα. Επίσης διαπιστώνουμε ότι τα δύο έγγραφα βρίσκονται σε διαφορετική φάση ζωής τους το παράδειγμα είναι ε, τελικό, ενώ η πρόταση της Κομισιόν στο αρχικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας ε, που θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο και το, ε, και το Κοινοβούλιο που μπορεί να μεταβάλουν την ουσία ή να εισάγουν κάποιο phasing in. Είναι πολύ νωρίς λοιπόν για να συγκρίνουμε τα δύο έγγραφα. Πολύ νωρίς για να το κατά πόσο αυτή η νομοθεσία θα καταστήσει το παράρτημα περιττό. Πιστεύουμε ότι είναι πολύ σημαντικό να δημοσιευθεί αυτό το παράρτημα τώρα και να εφαρμοστεί τώρα, διότι επιτρέπει την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Τα ξεκινήσαμε με τον ενιαίο αποπτικό μηχανισμό, οι τράπεζες, οι συνάδελφοι και ο φόρτος και μου έλεγαν ότι δεν, δεν έχουμε ανάπτυξη, περιμένετε μέχρι να έρθει ξανά η ανάπτυξη. Ναι, ε, ορίστε όμως η ανάπτυξη έχει έρθει εδώ και χρόνια, αλλά συνεχίζεται η παραγωγή κόκκινων δανείων. Και κατά τη διάρκεια αυτής της καλοήθους οικονομικής κατάστασης ξέρουμε πώς ε, δίνονται ε, κακά δάνεια, φτιάχνονται τα κακά δάνεια, όχι στην περίοδο κρίσης όπου όλοι πρόσεχαν και οι τράπεζες. Είναι καλή στιγμή τώρα λοιπόν ε, να ενεργήσουμε, να αναθεωρήσουμε να... τα κριτηριά μας ώστε να εξασφαλίσουμε ότι θα αντιμετωπιστούν ε, τα κόκκινα δάνεια από την αρχή, όπου δηλαδή είναι λιγότερο δυνηρό για τις τράπεζες, για τους δανειολήπτες και για την οικονομία. Αυτό σημαίνει παραγωγή περισσότερων δανείων. Όχι. Σύμφωνα με την έκτο και τις στατιστικές της, για τις οποίες δεν είμαι εγώ υπεύθυνη, αλλά είμαι βεβαία ότι είναι σωστές, έχουν πολύ καλή φήμη για τις ε, ε στατιστικές τους. Δεν βλέπω λοιπόν κανένα λόγο που θα έπρεπε να μας εμποδίσει να ενεργήσουμε τώρα. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα, υπάρχει κάποιο να μιλήσει από το ΕΛΚ, αν θέλετε. Ναι, ναι, ακριβώς. Εν τω μεταξύ, να δώσω τον λόγο στον κύριο Φερνάντες. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλώ ορίσατε και από πλευρά μου, κυρία Νουή. Μεγάλη μα χαρά που είστε εδώ. Εγώ θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Όπως γνωρίζετε, η κατάσταση των κόκκινων δανείων σε διάφορες δικαιοδοσίες εντό της Ένωσης είναι πρόβλημα για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε διάφορες ντοσχέ εντό τη ε, Τραπεζική Ένωση και μάλιστα χρησιμοποιείται για να αποφευθεί η πρόοδο σε ε, πολιτικά θέματα και σε διαπραγματεύσει. Τώρα θα ήθελα να σας ρωτήσω σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι τωρινές ε, συγκρίσεις ανάμεσα στα κόκκινα δάνεια διαφόρων χωρών είναι έγκυρες εφόσον ε, υπάρχουν πολλές διαφορές στα λογιστικά κριτήρια. Θα πρέπει να αξιολογήσουμε σε ποιο βαθμό αυτά τα ε, δάνεια είναι, ε, είναι σίγουρα. Δεν ξέρω λοιπόν ε, κατά πόσο αυτή η σύγκριση δίνει μια πιστή εικόνα της κατάστασης των διαφόρων τραπεζών εντός της, ε, Ένωσης, της Τραπεζικής Ένωσης. Η δεύτερη μου ερώτηση αφορά το γεγονός ότι ακόμα και αν ε, έχουμε προβλήματα όπως ας πούμε με την, την Banco Popular που έγινε πρόσφατα, με την με διάφορες τράπεζες. βάσει ε, περιπτώσει, στο πλαίσιο της αναθεώρησης, ε, της, ε, σε ποιο βαθμό μπορούμε να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία μας, ώστε αυτά τα, κρίσεις να μην καταλήγουν σε κρίσεις φεργιότητας. Το είπατε και εσείς, εξυγίανση, ρευστοποίηση, καθάριση. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε διάφορες χώρες. Ευχαριστώ πολύ. Thank uh, Σας ευχαριστώ πολύ. Ναι, τα μη να δάνεια είναι μεγάλο θέμα. Αλλά δεν είναι το μόνο θέμα προφανώς. Προφανώς πρέπει να απασχολήσει τις εποπτικές αρχές, αλλά και οι νομοθέτες πρέπει να λάβουν υπόψη τη μείωση του κινδύνου που αναπτύσσεται με την δημιουργία του ενίου εποπτικού μηχανισμού. Προφανώς θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαροι όροι για το σύστημα εγγύησης καταθέσεων και να μην χρησιμοποιούμε διάφορα προσχήματα. Νομίζω πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσουμε με αυτό το σύστημα και αν υπάρχουν κάποιοι όροι. Κατά την απόψή μας πρέπει να είναι καθορισμένοι εκ των προτέρων, να μπορούν να επαληθεύονται αντικειμενικά, να είναι ρεαλιστικά εφικτοί και να σχετίζονται νομικά με τις διάφορες φάσεις ε, του συστήματος εγγύησης καταθέσεων έτσι, ε, ώστε να μην αναβάλλεται αυτό επάπειρον το συντομότερο που θα, το συντομότερο, όσο συντομότερο να ξεκινήσουμε τόσο το καλύτερο. Και νομίζω ότι δημιουργείται τώρα μια νέα δυναμική για αυτό το ζήτημα. Για το θέμα είναι ακριβώς να φτάσουμε στην πλήρη αλληλεγγύη και το σύστημα εγγύησης καταθέσεων. Για την κρίση της ρευστότητας ε, υπάρχει πολύ ρευστότητα αυτή τη στιγμή στις ε, τράπεζες ε, και στην αγορά. Δεν υπάρχει έλλειψη ρευστότητας. Η ρευστότητα είναι το σύμπτωμα ότι κάτι δεν πάει καλά και αυτό δεν αλλάζει με μια αλλαγή κανονισμού που ούτως ή άλλως έχει αναπαθμιστεί με την μεταρρυθμίση, την τρίτη μεταρρυθμίση της Βασιλείας. Το θέμα είναι ότι το θέμα με τις τράπεζες είναι θέμα εμπιστοσύνης. Αν οι καταθέτες, οι καταναλωτές χάσουν την εμπιστοσύνη τους στις αγορές, τότε προφανώς υπάρχει μαζική ανάληψη καταθέσεων και ρευστού από τις τράπεζες ε, που δεν μπορεί να σταματήσει. Γι' αυτό η κρίση της ρευστότητας είναι ένα από τα στοιχεία που δείχνουν ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να αποφύγουμε το ότι ο πρώτος ο οποίος θα φτάνει συμβολικά στην πόρτα της τράπεζα είναι αυτός ο οποίος θα εξυπηρετείται πρώτος. Όταν αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις πρέπει να λάβουμε τέτοιε απότάσει Εκτός αν υπάρχει βεβαίω χρεοστάσιο που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, αλλά υπήρχε στην Λετωνία. Γι' αυτό ακριβώ ε, ε, ζητήσαμε τι εθνικέ αρχές να κάνουν κάτι τέτοιο, αλλά τότε η τράπεζα δεν μπορούσε να έχει ε, αρκετά γρήγορα επαρκή ρευστότητα για να πληρώσει τους ε, καταθέτες. Ε, είναι λοιπόν ένα δομικό πρόβλημα για τις τράπεζες. Αν χαθεί η εμπιστοσύνη τότε έχουμε πρόβλημα ρευστότητας, κάτι το οποίο βέβαιος ίσως έχει ξεκινήσει από ζητήματα ρευστότητας ή φερεγγιότητας. Τέλος πάντων, όταν χαθεί η φερεγγιοτητας παντων αυτό συμβαίνει. Μπρέαν Χέις. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε, καθώς πλησιάζουμε στο τέλος της ακρόασης. Όπως ε, θα ξέρετε τώρα έχουμε το φορολογικό πακέτο των ΙΠΑ που ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο και ένα κομμάτι είναι ένας ε, φόρος επαναποτρισμού 15% ε, που ενθαρρύνει τις πολυεθνικές να μεταφέρουν τα μετρητά τους από τις τράπεζες της Ευρωζώνης πίσω στις ΙΠΑ. Βεβαίω θα χρειαστεί ένα χρόνο να αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο αυτού. Έχετε κάποια ανησυχία για επαναπατρισμό καταθέσεων μεγάλη κλίμακας από τράπεζε τη Ευρωζώνης ε, προς τη ΣΥΠΑ από την σκοπιά του συστημικού κινδύνου ως ε, συνέπεια τέτοιου μαζικού επαναπατρισμού. δεν μπορώ να αξιολογήσω την κατάσταση σε αυτό το θέμα. Δεν ε, σχετίζεται ακριβώς με ρυθμιστικά ζητήματα, αλλά προφανώς εξετάζουμε όλα τα στοιχεία και θα δούμε αν υπάρχει λόγος ε, να αλλάξουμε άποψη στο προσεχές μέλλον για την ώρα, όχι πάντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα είναι η σειρά μου για την τελευταία ερώτηση. Και πάλι για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Τρία θέματα. Πρώτα είπατε δύο φορές και δείχνουν και τα στατιστικά σας στοιχεία ότι δεν έχουμε μία μείωση της πίστης. Δεν το αυτό, γιατί τα μέτρα δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα. Τι εννοείτε λοιπόν ε, με την αξιολόγησή σας αυτή. Και άκουσα και την κυρία τον να λέει ότι ο αντίκτυπος των νέων μέτρων θα είναι αμεληταίος ε, και διαχειρίσιμος. Αυτό ήταν μια υποκειμενική αξιολόγηση ή υπήρξε κάποια επιστημονική αξιολόγηση αντικτύπου. Υπήρχαν αριθμοί δηλαδή ήταν η άποψή της ή η δική σας άποψη. Γιατί είπατε ότι δεν υπάρχει ανάγκη αξιολόγηση αντικτύπου. Αμφιβάλλω γι' αυτό γιατί αυτά είναι μέτρα τα οποία θα επηρεάσουν συστηματικά τις ε, αρχέ. Πέρα από τους λογιστικούς κανόνες ε, και ειδικά στον πυλώνα 1. Είστε σίγουροι λοιπόν ότι δεν υπάρχει ανάγκη αξιολόγησης αντικτύπου. Δεύτερον, για την συμπληρωματικότητα. Άκουσα αυτό το οποίο λέτε ότι η πρόταση της Κομισιόν δεν έχει ακόμα εγκριθεί. Οπότε δεν ξέρουμε αν ήταν τελική. Κοιτάξτε, εγώ θα προτιμούσα μια ευθυγράμμιση εξ αρχής, αλλά τέλος πάντων ε, να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά όπως είπα και στην εισαγωγή μου, αυτή τη στιγμή ε, οριστικοποιηθεί η πρόταση της Κομισιόν. Έχω εδώ έναν πίνακα σύγκρισης, ε, παραδείγματος χάρη, μετά από 8 χρόνια ε, λέει η Κομισιόν ότι θα είναι τα ανοίγματα 40%, η Κομισιόν 70%. Μετά από την άλλη μεριά, σε ένα χρόνο η Κομισιόν λέει 35% μη ε, ασφαλισμένα, η Κομισιόν λέει 0%. Δηλαδή, μόλις ο πύλωνας ένα ενταχθεί στην ομοθεσία, έχει νόημα να έχουμε κάποιες οριζόντιες ρυθμιστικές προσδοκίες και πέρα από την ακόμα ανεπαρκή παροχή συγκεκριμένων τράπεζων για συγκεκριμένους λόγους. Και δεύτερον, έχει νόημα να έχουμε όχι μόνο οριζόντιες προσδοκίες, αλλά να είναι και διαφορετικές, να μην συμπίπτουν με αυτές τις νομοθεσίες. Και, και υπό τις δύο είναι καμιά φορά πιο αυστηρές, καμιά φορά λιγότερο αυστηρές. Τι γίνεται μετά, γιατί λέει ε, η Κομισιόν μετά από 7 χρόνια πρέπει να κάνετε αυτό και ο νόμος λέει πρέπει να κάνετε το άλλο. Εντάξει, τελικά θέλουμε να δούμε το τι θα ποια θα είναι η τελική μεταρρυθμίση, εντάξει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάποια ευθυγράμμιση, αλλιώς δημιουργείται σύγχυση. Τρίτον, η Κομισιόν κάνει μια διάκριση μεταξύ του ε, απίθανο να πληρωθεί και ε, πέραν της προθεσμίας. Γιατί ε, δεν έκανε κάτι τέτοιο η δική σας αρχή. Από την άλλη βλέπουμε ότι γίνεται μία διάκριση η οποία αφορά κάτι το οποίο αναφέρεται ως τρέχουσες και διαρκείς ε, ανησυχίες για τα εκπρόθεσμα δάνεια. Οπότε, από αυτήν την έννοια, η αξιολόγηση δική σας είναι μάλλον καλύτερη. Τι άποψη έχετε ακριβώς για το ότι η Κομισιόν δεν κάνει αυτή την διάκριση στην πρότασή τη Και τέλος, για τις εγγύησει, λέτε ότι τελικά θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα ανάκτηση ε, τη εγγύηση. Ξέρετε πως ε, υπάρχει και υπάρχουν και διαφορετικές νομικές διαδικασίες και θυμάμαι στο έγγραφο του Συμβουλίου υπήρχε μια πρόταση για να γίνει μια διάκριση όταν υπάρχει, να υπάρχει μια εξωτερική ανεξάρτητη αξιολόγηση για το αν έχει κάποια αξία ακόμα η εγγύηση. Γιατί λοιπόν μιλάμε για το μηδέν ε, Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ας πούμε κάτι το οποίο όντω έχει μηδενική αξία, αλλά μπορεί να υπάρχει ένα μέγαρο το οποίο θα έχει όντως ε, αξία. Δεν ξέρω γιατί επιμένετε στο, στη μηδενική αξία. Στην Κομισιόν ε, κατά κανόνα δεν ισχύει αυτό. Ίσως και αυτός είναι ένας άλλος τομέας όπου πρέπει να υπάρξει κάποια βελτίωση. Ευχαριστώ. Πολλά ξεχωριστά σημεία. Όταν σας είπα δεν υπάρχει περιορισμός της χορήγησης ε, δανείων, εννοούσα ότι ε, εξετάζουμε διαρκώς την ε, τροφοδοσία με δάνεια και βλέπουμε ότι όλα είναι εντάξει, δεν μειώθηκαν δηλαδή τα δάνεια ε, λόγω του παραρτήματος. Όταν τώρα μιλάμε για την αξιολόγηση αντικτύπου, όταν ε, μιλάμε για αντικειμενικά και επιστημονικά στοιχεία, Ξέρετε, είναι μεγάλη ψαλίδα ανάμεσα ε, στα επιστημονικά και στα αντικειμενικά στοιχεία. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ε, εναλλακτικές λύσεις με διάφορο βαθμό, διαφορετικό βαθμό αξιοπιστίας. Ξέρετε ότι διάφορα μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου και ενίοτε και με σύγκρουση συμφερόντων έχουν εκπονήσει εκτιμήσεις και κάποιοι θεώρησαν ότι δεν ήταν σωστά τα στοιχεία, ε, άλλες αναλύσεις αποκλίναν από τις προηγούμενες. Σε κάθε περίπτωση, για τις εκθέσεις ε, σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια, είδαμε στο παράρτημα ότι ήταν ε, όχι αμελητό, αλλά διαχειρίσιμο το ποσό. Οπότε χρησιμο... εμείς βασιστήκαμε σε εμπειρικά δεδομένα και αυτό απέδειξε ότι δεν χρειαζόμασταν άλλη αξιολόγηση αντικτύπου. Όταν ε, όμως ε, μιλάμε για τα αποθέματα, άλλο καπέλο αυτό θα χρειαστεί άλλη μελέτη αντικτύπου. Υπάρχουν διαφορές ανάμεσα ε, στα όργανα του πυλώνα 1 και του πυλώνα 2. Ναι, αλλά αυτό είναι και η λογική του πυλώνα 2. Η νομοθεσία σχετικά σχετίζεται με τον κίνδυνο σε τράπεζα μεσαίου μεγέθους. Και από αυτή την άποψη είναι μεγαλύτερο αυτός ο κίνδυνος από τον μεσαίο κίνδυνο και άρα οι εποπτικές αρχές θα πρέπει να επιληφθούν. Ρωτάτε τι πρέπει να κάνει η τράπεζα, μα να συμμορφωθεί με τον κανονισμό, αρχίζοντας με τον πυλώνα 1. Πρέπει να συμμορφωθεί ασυζητητή και μετά. Θα δούμε τι πρέπει να γίνει μέσα του υποπτικού διαλόγου, με, πέρα από τον πυλώνα ένα, δηλαδή θα αποδείξουμε στην τράπεζα ότι ο κίνδυνός της επερβαίνει το μέσο όρο για την αφηγία ή για οτιδήποτε άλλο, διότι το κανονιστικό πλαίσιο της χώρας ε, δεν λειτουργεί καλά για την επανάκτηση εγγυήσεων και ούτω καθεξής. Οπότε ναι, απαντοκαταφατικά πάντοτε θα υφίστανται διαφορές ανάμεσα στους δύο πυλώνες και όχι μόνο για την έκθεση στα κόκκινα. Διακόπτει ο κ. Γκουαλτιάρη. Λέτε ότι το μέσο όρο είναι στα πυλώνα 1. Και μετά λέει μία τράπεζα μπορεί να έχει την τα αναφύγικα... Οπότε και αυτό μέσος κίνδυνος δεν είναι. Ποιο, νόημα να έχουμε τους δύο πυλώνες. Κοιτάξτε, δεν είναι τώρα το σωστό χρονικό σημείο για να κάνουμε οποιαδήποτε σύγκριση. Όταν και εφόσον ο πυλώνας να έχει ως αποτέλεσμα να είναι περιττό ε, το παράρτημα, ας γυρίσουμε τη σελίδα και ας κάνουμε κάτι άλλο. Αλλά εγώ πολύ αμφιβάλλω. Εγώ πρώτη θα πετάξω τη σκούφια μου, άμα συμβεί αυτό. Πολλά θα γίνουν μέσα από το IFRS 9, γιατί σε σχέση με το IES 39 είναι υψηλότερε οι υποχρεώσεις και θα καλύπτουμε τις πραγματικές απώλειες ε, και όχι μόνο τις δεδουλευμένες. Οπότε ο, το περιθώριο θα είναι πολύ μικρότερο για τον πυλώνα 1 σε σχέση με τον πυλώνα 2. Μήπως εκ, εκλείψει, γιατί θα είναι τόσο μικρό το περιθώριο, δεν το ξέρω όμω αυτό. Σε κάθε περίπτωση θα είναι μικρότερο. Πάντως διαφοροποίηση θα έχουμε κάνει, διότι δεν πρόκειται για νομικές διατάξεις, ε, πρόκειται για μια συζήτηση για εικασίες, ίσως με την, ε, από τη συζήτηση προκύπτει, ε, προκύψει ότι δεν χρειάζεται. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Για την αξία των εγγύσεων με ρωτήσατε, αν αυτό την επηρεάζει. Μα όχι. Ζητάνε εγγύηση για τη δανειοδοσία η τράπεζες διότι θέλουν μια δικλίδα ασφαλείας, οπότε πρέπει να είναι και σε θέση να επανακτήσουν την εγγύηση μετά την πάροδο κάποιου αριθμού κάποιων ετών, εάν δεν αποπληρώνονται τα δάνεια. Μπορεί να είναι εξαιρετικά υψηλή η αξία, όμως εάν δεν είναι δυνατή η επανάκτηση, δεν έχει και κανένα νόημα. Όποια και αν είναι η αξία της εγγύησης, χαμηλή ή υψηλή. Εδώ μιλάμε για υποστηριζόμενο από, τις, ε, από εγγύησεις ε, δάνειο και εκπνέει αυτή η εγγύηση, άσχετο τι αξία έχει μετά από την πάροδο κάποιων ετών. Δεν είναι το βασικό μας ζήτημα ε, το ύψος των εγγύησεων. Γουαλτιέρη. Ευχαριστούμε. Πιστεύω ότι ήταν πολύ χρήσιμος αυτός ο διάλογος και είπατε ότι από τον πυλόν ένα μπορεί τελικά να εκλειψεί και η ανάγκη για το παράρτημα. Θεωρώ ότι είναι θετικό αυτό που είπατε και μπορεί οι νομοθέτες να το εκλάβουν ω ενθαρρυντικό στοιχείο για να επισπεύσουν. Αλλά μπορεί ταυτόχρονα να γυρίσει και μπούμεραν αυτό που είπατε. αλλά σε κάθε περίπτωση ε, δεν μπορείτε εσείς να προδικάσετε την έκβαση. Αν είναι υγιές το σύστημα πυλώνα 1, Δεν χρειάζεται να μιλάμε για συγκεκριμένο αριθμό ετών, διότι θα μιλάμε για τον πυλώνα 2 και την, την, τη μη επαρκή ε, παρουσία στοιχείων ενεργητικού. Για το ξέπλυμα χρήματος, όπως είπε και ο Γκίγκολτ, εσείς είσαστε υπέρ της εναρμόνισης Λοιπόν, θα, θα ε, αξιολογήσουμε όλες τις εναλλακτικέ λύσεις ε, και το ε, SSM, ο νέος εμποπτικός μηχανισμός, θα, θα μετέλθει όλων των διαθέσιμων μέσων για να μπορέσουμε Έχουμε ένα business model για την, το, την καταπολέμηση της νομοποίησης χρημάτων από παράνομες δραστηριότητες. Σας ευχαριστούμε. Colleagues, before I pass the chair to uh, uh, Αδελφοί, πριν δώσω την προεδρία στον Μάρκους, να σα ενημερώσω ότι λόγω απεργιών σε Γαλλία και Βέλγιο αύριο το πρωί, ο Επιτροπός Μοσκοβισή ζήτησε να καθυστερήσει η έναρξη της συνεδρίασης κατά 15 λεπτά. Οπότε θα ξεκινήσουμε 9 και 4. Έτσι, ένα προληπτικό περιθώριο, θα έλεγα, μια προληπτική διάταξη. Από αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία ε, ελπίζω να μπορέσουμε εμείς να είμαστε όλοι εδώ εγκαίρους γιατί η απεργία μας αφορά όλους, όχι μόνο τον Επίτροπο. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, βιώσιμη χρηματοδότηση, δίνω τον λόγο κατευθείαν στην εισηγήτρια, την Μόλι Σκοτ Κέιτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ ε, που προφέρατε και το όνομά μου σωστά. Σας ευχαριστώ. Τώρα πλέον το θέμα έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης της ε, ε, των αρχών. Είχαμε τον Γάλλο Πρόεδρο και δύο επιτρόπους την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε βλέπετε ότι έχει φτάσει και στους ανώτατους όροφους ε, της ε, Κομισιόν αλλά και τα υψηλότερα επίπεδα. Είναι λοιπόν πολύ ενθαρρυντικό, υπάρχει θα έλεγα πολιτική συμφωνία όλων των ομάδων. Καταφέραμε να παραμερίσουμε τις πολιτικές διαφωνίες μας γιατί όλοι συμφωνούμε για την ανάγκη να ανταποκριθούμε στην κλιματική κρίση και να μετακινηθεί εκεί πέρα η χρηματοδότηση, κάτι το οποίο ξεπερνά τις άλλες πολιτικές μας διαφωνίες. Και οπωσδήποτε αυτό συνέβη και με τους κοιόδες εισηγητές μου και εκτιμώ ιδιαίτερος ε, το πόσο ε, βοήθησαν με τις ε, τροπολογίες τους, τις οποίες επέβαλαν με θετικό πνεύμα θα έλεγα. Ήδη είχαμε μια συνάντηση των σχεδόν εισηγητών που αποτέλεσε νομίζω μια καλή βάση και για το μέλλον. Τα ζητήματα τα οποία θα καλύψουμε περιλαμβάνουν αποκάλυψη, είπε η πράσινη χρήματα αγορά, και τα σχετικά και θα ήθελα και εγώ βεβαίως να πω πως το Κοινοβούλιο δεσμεύεται ε, για κάτι τέτοιο. Συμφωνήσαμε λοιπόν για τη σημασία της υποχρεωτικής αποκάλυψης ε, τέτοιων στοιχείων του ενεργητικού τα οποία δεν είναι βιώσιμα. Μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν μεγάλες ε, διαφωνίες, αλλά αντιλαμβάνομαι ότι συμφωνούν οι περισσότερες ομάδες. Επίσης είπαμε ότι θα πρέπει τα καθήκοντα προς τις ε, εταιρείε ε, της διοίκησης θα περιλαμβάνουν και τέτοια ε, τέτοια είδου πληροφορίε που θα φτάνουν μέχρι και την αλυσίδα των προμηθευτών. Μέχρι στιγμή δεν έχουμε καταλήξει στην ανάγκη για το πώς θα μετρήσουμε τέτοιες ανάγκες κεφαλαιοποίησης. Συμφωνούμε στο ότι θα πρέπει να μειωθούν ε, οι, τα τέτοια στοιχεία ενεργητικού τα οποία παραμένουν ε, και είναι μη βιώσιμα αλλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα πώς θα γίνει αυτή η μετάβαση. Όσον αφορά τον πράσινη, τα ξονομία των πράσινων ομολόγων. Ελπίζουμε να συνεισφέρουμε σε κάτι χρήσιμο. Συμφωνούμε για την σημασία μιας πανευρωπαϊκής ομάδας ε, των ενδιαφερομένων ε, για τα στοιχεία εκείνα τα οποία θα αφορούν τις μη χρηματοοικονομικές ε, αναφορές και εντός του Κοινοβουλίου ελπίζουμε να επιτύχουμε μια ευρεία συμφωνία ταξονομίας η οποία θα βασίζεται σε δείκτες που υπάρχουν ήδη ε, που αφορά το οικολογικό κόστος ε, και όφελος ε, του πλανήτη και να επιτρέψουμε έναν ορισμό του βιώσιμο ο οποίος θα είναι ουδέτερος τεχνολογικά. Και θέλουμε βεβαίω να τοποθετηθεί και το Κοινοβούλιο με τρόπο που θα μπορέσει να καθοδηγήσει και τη δουλειά της ομάδας των ενδιαφερομένων. Επίσης θα πρέπει να δούμε τα συνταξιοδοτικά προϊόντα μέσω μιας νομοθετικής πρωτοβουλίας και ενιαίας ε, διατάξεις για τα πράσινα ομόλογα. Θεωρούμε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι διακριτά από το να περάσουν οι επενδύσεις ε, στην πράσινη κατεύθυνση. Γιατί βεβαίω δεν έχει πάρα πολύ νόημα αν δεν φύγουν τα λεφτά από τις μη βιώσιμες επενδύσεις. Είμαστε πεπισμένοι, τουλάχιστον εγώ είμαι πεπισμένοι ότι δεν θα πρέπει να περιλαμβάνουν ορυκτά καύσιμα, αλλά εμείς θα θέλαμε να αποκλειστούν επίσης και οι αερομεταφορές και η πυρηνική ενέργεια. Και ανησυχούμε για το ότι θα πρέπει οι παράγοντες αυτοί να περιληφθούν στις αξιολογήσεις των οίκων αξιολόγησης για να υπάρξει μια σοβαρή εφαρμογή αυτών των προδιαγραφών και μια διαδικασία πιστοποίησης ε, των πράσινων επενδύσεων, ε, πιθανότατα υπό την εποπτεία της ΕΣΜΑ. Τέλος, θα πρέπει ακριβώς ε, να δώσουμε και εμείς το καλό παράδειγμα και ε, δεν μπορούμε να περιμένουμε οι επενδύσεις να πάνε προς αυτήν την κατεύθυνση εάν ε, τα δικά μας τα θεσμικά όργανα επενδύουν σε μη βιώσιμα στοιχεία Μιλάω εδώ πέρα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ότι θα πρέπει ακριβώς να δούμε τις θεσμικές ελλείψεις που υπάρχουν σε αυτόν τον ε, τομέα. Βλέπουμε ακριβώς ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε υψηλό επίπεδο. Είχα κάποιες συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά δυστυχώ πρόσφατα επένδυσαν 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ στον αγωγό της ε, Ανατολής που μας δεσμεύει για πολλές δεκαετίες και πρέπει ακριβώς να αλλάξουμε και την εντολή της ΕΝΙΖΑ για να περιλαμβάνει και τους σχετικούς κινδύνους και να ευθυγραμμιστεί με την Συμφωνία των Παρισίων και τους σχετικούς στόχους και να φροντίσουμε να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους και να υπάρχει και ακριβώ μια συνέπεια με τους στόχους περί κλιματικής αποκάλυψης. Πολλές και συναρπαστικές τεχνικές λεπτομέρειες, μέχρι στιγμής η πρόοδος είναι πάρα πολύ καλή και ευχαριστώ και τους ε, σκιώδεις εισηγητές και αναμένω τις ε, περαιτέρω συζητήσεις. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έρχομαι λοιπόν τώρα στους σκιώδεις εισηγητές. Ξεκινάμε με το ΕΛΚ. Ο Μπράιν Χέιζ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, εξ ονόματος ε, των, της κυρίας Πιετικάινεν θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και τους και οδησηγητές για την πολύ επικοδομητική συζήτηση που είχαμε για το θέμα αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι το σχέδιο έκθεσης πηγαίνει προς την σωστή κατεύθυνση για να δημιουργήσει ένα κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Θα αποστείλει ένα σημαντικό μήνυμα για, για την θέση του Κοινοβουλίου ε, προς τα κράτη μελη εν ώψη του σχεδίου δράσης. Το σχέδιο έκθεσης ε, κάνει κάποια καλά βήματα προς την διασφάλιση ενός ρυθμιστικού πλαισίου που θα δίνει κίνητρα για να προχωρήσει η μετάβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς μια βιώσιμη οικονομία σύμφωνα με τους στόχους των Παρισίων. Τα μέτρα για να διορθωθούν οι τωρινές αποτυχίες της αόρας βεβαίως είναι ευπρόσδεκτα. Υπάρχουν κάποια στοιχεία όμως τα οποία απαιτούν περαιτέρω συζητήσει και τα οποία θα γνωρίζει η συγγήτρια. Πρώτα απ' όλα οι απαιτήσει θα πρέπει να είναι οι καταλληλές και να είναι αναλογικές όσον αφορά το μέγεθος ε, των επιχειρήσεων και τους κινδύνους που αντιμετωπίζει. Οι νέες απαιτήσει δηλαδή θα πρέπει να δημιουργήσουν δυσανάλογο βάρος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δεύτερον, οποιαδήποτε προληπτική αντιμετώπιση των μη βιώσιμων στοιχείων ενεργητικού θα πρέπει να μην δημιουργήσει ένα μηχανισμό στρέβλωσης της αγοράς που θα ενθαρρύνει την ανάληψη κινδύνων που θα οδηγήσουν σε φούσκες και περαιτέρω κινδύνου στο μέλλον. Τρίτον και σημαντικότερον πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί όταν μιλάμε για την μελλοντική ε, ταξονομία ή το πράσινο σήμα. Για να αξίζει κάτι τέτοιο θα πρέπει να βασίζεται σε δείκτες βιωσιμότητας, ε, μετρήσεις και να αποκαλύπτει τον αντίκτυπο στο περιβάλλον και στο κλίμα αντί να οδηγεί σε κάτι το οποίο απλά θα κάνουν οι επιχειρήσεις ως ε, γραφειοκρατία για την μέτρηση των εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα, αποτελεσματική χρήση πόρων, κατανάλωση υδάτων, βιοπικιλότητα, παραγωγή απορριμμάτων, μεταξύ πολλών Υπάρχουν ήδη και αναπτύσσονται τέτοιοι δείκτες από διάφορες αρχές, την Κομισιόν, τον ΟΣΑ, τον ΟΗΕ και τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει τώρα είναι να υπάρξει μια εναρμόνιση των δικτών ε, που χρησιμοποιούν οι εταιρείε. Ευχαριστούμε λοιπόν ιδιαίτερο την εισηγήτρια για την ε, συνεργασία. να Αναμένουμε την συνεργασία μας ε, με σκόπο ένα στιβαρό ρυθμιστικό πλαίσιο που θα δώσει δυνατότητα σε όλους τους εμπλεκόμενους να δραστηριοποιηθούν σωστά. Σοσιαλιστές η Ευχαριστούμε. Ε, ελπίζω και η Σιμώνα Μποναφέ να έρθει από την ομάδα μας. Για κάποιες τροπολογίες θέλω να κάνω σχόλια για να αποφύγουμε αυτά τα τεστ κοπόσεως ε, σε σχέση που γίνονται σε σχέση με τις συστάσεις ε, της ΕΚΤΕ, τροπολογία 100. Στο μακροπροληπτικό πλαίσιο πρέπει να ενσωματώσουμε τον κίνδυνο. που Χρειαζόμαστε add-on ε, σε, όπως περιγράφουμε στις 163, 165 και 166. Επίσης, ε, ε, βαλτιστές πρακτικές από την εθνική νομοθεσία για την αποκάλυψη πληροφοριών, άρθρο 173 της ενεργειακής νομοθεσίας και θα πρέπει λοιπόν για την ιδέουσα επιμελητή να αναφερόμαστε σε τέτοια ε, είδη εθνικής νομοθεσίας. Ε, ε, τρίτον, για την αξιονομία πιστεύουμε ότι πέρα από τη, την πράσινη διάσταση θα πρέπει και να είναι εξίσου ενισχυμένη και η κοινωνική διάσταση και η διάσταση της διακυβέρνησης. Μην ξεχνάμε τις ε, μη αναμενόμενες επιπτώσεις που είχαμε μέχρι στιγμής ε, για τους νέους κινδύνους κυρίως, ε, για το πλαίσιο ε, χρειαζόμαστε και κοινωνική διάσταση, ε, πρώτερη συγκατάθεση από τις ε, τοπικές κοινότητες όταν επηρεάζονται και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πέμπτο σημείο, χρειάζεται η ταξονομία αλλά δεν επαρκεί είναι, έχει σημασία, πάρα πολύ μεγάλη σημασία η υποχρεωτική ταξονομία για τον ε, εντοπισμό και την πρόληψη των κινδύνων από πλευρά ε, κοινωνική, οικονομική και διακυβέρνηση ε, και γι' αυτό προτείνουμε τι τροπολίε 110 και 114. Το θέμα των πράσινων ομολόγων προτείνουμε ε, την ε, τροπολογία 230. έκτη παρατήρηση. Ε, σε όλη την ε, επενδυτική αλυσίδα θα πρέπει να έχουμε υλικούς παράγοντες EST τροπολογία 201 δηλαδή νομοθετικό πλαίσιο για την έκδοση υπερσυνομολόγων από ε, τρέχοντα και μελλοντικά ιδρύματα, τροπολογία 230, όπως σας έλεγα προηγουμένως. Και τέλος, η δομή θα πρέπει να περιγράφεται ε, όπως στις τροπολογίες 287 και 303 και ελπίζουμε να είναι καλή η συνεργασία μας, ε, αλλά από ό,τι φαίνεται θα είναι όπως έχουμε δει μέχρι στιγμής. Ευχαριστούμε. ECR, μπορείτε να σβήσετε το, το μικρόφωνο σας, πύρκο. Ευχαριστώ. Πάρα πολύ καλή συνεργασία μας, ε, γιατί είναι και εξαιρετικά περίπλοκο το θέμα. Ο στόχος είναι τα κριτήρια ESG, οικονομικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης, να ενσωματωθούν σε όλες τις μορφές μιας βιώσιμης βιοοικονομίας. Είναι μεγάλη η πρόκληση Ταυτόχρονα πρέπει να ε, λάβουμε υπόψη τις πολλαπλές ε, αποτυχίες ε, της αγοράς, το εξωτερικό περιβάλλον, τη μόλυνση, τον συστημικό κίνδυνο στις κεφαλαιαγορές και αυτό απειλεί την σταθερότητα της οικονομίας. Εγώ τονίζω πως δεν πρέπει να έχουμε ευρωομόλογα για το πράσινο ξέπλυμα ή ε, αποδυναμωμένη ε, διακύβευση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή οικονομικής ε, αστάθειας. Οι λύσεις μου βασίζονται στην αγορά. Να σταματήσουμε την έκδοση των αδειών χωρίς έλεγχο και απλέ, απλ, ε, απλούστευση της υποβολής εκθέσεων. Ε, πιστεύω ότι πρέπει να είναι ξεκάθαροι οι κανόνες για τη νέα ταξινομία και για άλλα συναφή ε, νομοτεχνικά ζητήματα, τους ώστε στην πράξη να εφαρμοστούν ευκολότερα και να αποφύγουμε κόστος και χρόνο που μπορούμε να εξοικονομήσουμε. Ε, στατιστικά στοιχεία χρειαζόμαστε, αλλά φυσικά θα πρέπει να είναι ε, όσο τον πιο συγκρίσιμα γίνεται. Και μπορούμε να κάνουμε προσπάθειες με τους ε, ε άλλους σκιώτες εισηγητές να καταλήξουμε σε κοινώς αποδεκτές συμβαστικές λύσεις. Ευχαριστώ. Η Λιέβη για τους φιλελευθέρους. Λιέβη Βίρινγκ, ευχαριστώ. Αγαπητή συγγήτρια, αγαπητοί συνάδελφοι. Με ικανοποιούν οι ιδέες που αποτυπώνονται στις τροπολογίες ε, για τις έκθεσεις ε, με κριτήρια ESG ε, οικονομικά, κοινωνικά και διακυβέρνηση. Έχουμε αλληλοσυμπληρώμενου στόχους. Τι θέλουμε όλοι, να πάνε τα χρήματα σε πιο βιώσιμε επενδύσει. Για να ενισχύσουμε την βιωσιμότητα των ε, ε, χρηματοπιστωτικών αγορών. Καλωσορίζουμε τις προσπάθειες που έχουν γίνει για να γίνει βιωσιμότερη η οικονομία και θα πρέπει να συνεχίσουμε να τις υποστηρίζουμε. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν θέλουμε να καλύψουμε το επενδυτικό χάσμα και να επιτύχουμε τους στόχους μας, πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Πρέπει να, όχι μόνο να αμείβουμε αυτούς που είναι ήδη βιώσιμοι, ε, να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις που πρέπει να κάνουν τη μετάβαση. Πρέπει και εκείνες να έχουν τα μέσα για να το κάνουν. Και σε ένα σταθερό περιβάλλον, ναι, με τακτικό τρόπο. Φυσικά χρειάζονται αλλαγές στην πολιτική για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Όμως δεν πιστεύω ότι η νομισματική πολιτική είναι το σωστό εργαλείο. Για μένα είναι δύο τα στοιχεία κλειδιά που πρέπει να ε, μας απασχολήσουν περισσότερο. Ε, να είναι περισσότερε οι πληροφορίε διαθέσιμε για να, γίνουν, να λαμβάνουν σωστέ επενδυτικέ αποφάσει και τα εργαλεία αυτέ οι αποφάσει ε, να ε, μπορούν να μετατρέπονται σε συγκρίσιμου δείκτε. Αυτό δεν αντικαθιστά απέκτηση τη αγορά. ούτε τροποποιεί του κανόνε ενισχύουν την ικανότητα που έχουμε και που έχουν επιχειρήσεις να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους. Ταυτόχρονα θα πρέπει να μεριμνήσουμε ώστε η αποκάλυψη πληροφοριών να περιοριστεί στις πιο χρήσιμες και σημαντικές πληροφορίες. Πρέπει να υπάρχουν ξεκάθαρα κατόφλια για να μην έχουμε μεγάλο διοικητικό άχθος για τις επιχειρήσεις για την ταξινομία. Δεν είναι ο στόχος μας τώρα να προσδιορίσουμε ούτε τη δομή ούτε το περιεχόμενό της. Τη διακυβέρνηση αυτό πρέπει να αποφασίσουμε το ώστε να έχουμε το ευκταίο επίπεδο αντικειμενικότητας αλλά και ε, χρηματοπιστωτικής και τεχνικής επιρρογνωμοσύνης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα για όλους μας και γι' αυτό θα ήθελα να επικεντρωθούμε όλοι στην ουσία της συζήτησης. Σας ευχαριστούμε. Δεν βλέπω κανέναν από την ΚΟΕ. Ε, ωραία, να πάμε στο Catch the Ποιος θέλει το λόγο. Κανείς. Ορίστε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω την ε, εισηγήτρια για το εργασία της. Έχουμε ενώπιον μας ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας επιτρέπει να ε, επιτύχουμε τους στόχους του Παρισιού και να προχωρήσουμε προς ένα πιο βιώσιμο σύστημα. Πρόκειται για μια μετάβαση που σημαίνει πολλές επενδύσεις, ε, πολλά εκατομμύρια στο πλαίσιο ενέργεια και περιβάλλον. Δεν μπορούν αυτά να ε, δοθούν όλα αυτά από το δημόσιο τομέα, κανένα κράτου, οπότε βασικά θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από τον ιδιωτικό ε, τομέα. Ήδη υποβάλαμε διάφορε τροπολογίε, τι ε, ανέφερε και η συνάδελφο Μπερέ, που αφορά τι ισχύουσε νομοθεσίε. Η πρόκληση είναι πολύ μεγάλη και περιμένουμε από την Κομισιόν και νέε νομοθετικέ προτάσει, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε κι εμεί τον νομοθετικό μας ρόλο. Ε, εξάλλου είναι ακόμα πιο σημαντικό μετά τις 8 Μαρτίου και τη δημοσίευση του σχέδιου δράσης ε, της ε, Κομισιόν. Οι προτάσεις που έχουν ανακοινωθεί με βάση αυτή της ταξονόμησης σημαίνει, ε, σημαίνουν ότι θα είναι περισσότεροι ε, ε, μεγάλες και σημαντικές για την Ευρώπη. Τι είναι βιώσιμο και τι όχι όσον αφορά την ε, ταξονομία. Ε, θα πρέπει να, όλα αυτά να βασιστούν στην ε, διαφάνεια. Η 147 τροπολογία αφορά αυτό το θέμα. Όλα τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα θα πρέπει να, ε, ε, ανταποκρίνονται στα κριτήρια τα περιβαλλοντικά και της διακυβέρνησης. Επίσης, οι μεμονωμένοι υποταμευτές θα πρέπει να έχουν ενημέρωση όσον αφορά τον περιβαλλοντικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο των επενδυτικών τους επιλογών. Επίσης, ε, δεν θέλουμε να μιλήσουμε μόνο για τα κανόνες χωρίς να δούμε τα χαρακτηριστικά του βιομηχανικού ιστού που θα πρέπει να ε, στηρίξει τη μετάβαση. 180 δις ε, επενδύσεων το χρόνο στην ενέργεια έχουμε υπολογιστεί. Για το θέμα της πάυσης χρήσης του άνθρακα εντάσσεται και η 155 της αποτελεσματικής χρήσης δηλαδή των πόρων, το ε, παράγοντες ανταγωνιστικότητες δηλαδή μιας οικονομίας δεδομένης ε, της περατής φύσης των πόρων. Ε, έχουν ήδη μελετηθεί όλα αυτά ε, και σημαίνει εκβάθρον ε, αναθεώρηση του βιομηχανικού μας ιστού. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να ορίσουμε την θέση μας με αυτό το έγγραφο για τη βιώσιμη οικονομία. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι οι κανόνες θα πρέπει να απλοποιούν και να διευκολύνουν τις δυνατότητες ε, των βιομηχανιών για να μπορέσουν δηλαδή να ζητήσουν τα απαραίτητα, τις απαραίτητες πιστώσεις. Οι κίνδυνοι είναι με, ε, αρκετά μεγάλη αν δούμε όμως ε, με το μέσο και το μάκρο πρόθεσμο ορίζοντα μειώνονται και βεβαίω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τα κριτήρια, τα προληπτικά και λαμβάνοντας υπόψη και το, το μέγεθος των επενδύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Σιμώνα. Δεν έχω άλλον στον κατάλογο, οπότε θα ζητήσω, α, από την Μόλι να συνοψίσει. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ε, συμφωνώ καταρχάς με το όσα είπε η Λέιβε που είπε ότι είναι πολύ σημαντικό που πρώτη φορά έρχεται ένα τέτοιο θέμα στο Κοινοβούλιο και θέλω να σας παροτρύνω να λάβετε υπόψη όλα αυτά τα θέματα γιατί υπάρχουν ε, αλληλένδετα ε, ζητήματα που διέπουν πολλούς από τους φακέλους που μας απασχολούν εδώ. Θα πρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα και πολιτική κατεύθυνση από τους συναδέλφους εδώ και από την Κομισιόν και από ό,τι κατάλαβα η Κομισιόν, το Συμβούλιο είναι ευνοϊκό προς κάποιες από αυτές τις προτάσεις. Έχουμε λοιπόν ευνοϊκό άνεμο, ούριο άνεμο και θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε σχετικά σύντομα από ό,τι φαίνεται. Άκουσα τα σχόλια κάποιων σκιωδών για το πόσο σημαντικό είναι να συμπεριληφθούν ευρύτεροι ε, στόχοι της χιλιετίας ε, αλλά για να γίνει ένα επιτυχές κείμενο και να συνταχθεί μια νομοθεσία που να μπορεί να εφαρμοστεί, πρέπει να έχουμε λεπτομέρειες για το ποιους δείκτες πρέπει να έχουμε. Πρέπει να έχουμε μετρήσιμες ιδέες. Οπότε αυτές αναζητώ. Ε, διαφορετικά θα πρέπει να τα βάλουμε αργότερα εδώ. ο κίνδυνος ο περιβαλλοντικό είναι ο πιο πιεστικό, αλλά υπάρχουν και ένα σωρό άλλα ζητήματα που προέρχονται από την ευρύτερη οικολογική κρίση. Ε, σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλιά σας και ε, προσβλέπω στη συνεργα... μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Το χρονοδιάγραμμα, όπως σας έχω ήδη ανακοινώσει, ισχύει και προβλέπεται η ψηφοφορία στη συνεδρίασή μας στα τέλη Απριλίου μπορέσετε να διπραγματευτείτε μέχρι τότε. Πριν να περάσουμε στο σημείο 5, θα δώσω την προεδρία στον συντονιστή των σοσιαλιστών, στην συντονιστή των σοσιαλιστών, την Περβάνος Μπέρες.

τους ε, βουλευτές ε, και την εισηγήτρια. Ξεκινάμε την συζήτηση για το θέμα 5, έλεγχος των κατεξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών μέτρων. Σημερινό θέμα είναι η οδηγία και κεφαλαίων απαιτήσεων 4. Έχουμε λοιπόν την 36η τέτοια συνεδρίασή μας. Όπως γνωρίζετε αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην αποτελεσματική άσκηση των ε, αρμοδιοτήτων μας αυτών θεωρούμε ότι μία δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα είναι ο καλύτερος τρόπος για να ασκήσουμε αυτές τις αρμοδιότητες και σήμερα βεβαίως θα ασχοληθούμε με αυτές τις, την οδηγία και τον κανονισμό περί κεφαλιακών απαιτήσεων που αποτελούν τον πυρήνα της σχετικής νομοθεσίας για την ώρα. Περιέχουν εξουδότηση προς την Κομισιόν για να προβεί σε πράξεις ε, κάθε εξουσιοδότηση για να εφαρμόσει τεχνικές ε, προδιαγραφές που βασίζονται σε κάποια σχέδια τα οποία έχει επεξεργαστεί η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Αυτά τέθησαν ισχύ το 2014 και έχουμε ήδη και αρκετή δευτερογενή νομοθεσία, όμως ε, κρεμούν ακόμα, ε, κρεμούσαν ε, τον Φεβρουάριο αρκετά νομοθετήματα τον Ιανουάριο πέρσι. Εν μεταξύ έχουν εγκριθεί πολλές πράξεις κατά εξοδότηση, δύο ακόμα έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν και είναι υπό την έξεταση του Κοινοβουλίου, πέντε άλλες τέτοιε ε, έχουν αποτελέσει αντικείμενο σχέδιου γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής ε, Τραπεζικής Αρχής και αναμένουμε την ειδοποίηση της Κομισιόν καθώς σύμφωνα με το άρθρο 10 έχει η Κομισιόν τρεις μήνες να αντιδράσει. Αυτό σημαίνει όμως ότι έχουμε ακόμα 11 πράξεις κατεξοδότηση. Σύμφωνα με το άρθρο 460 που έκρεμει ακόμα και σημειώνουμε έτσι το ότι το 2015 και 2016 η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή ζήτησε από την Κομισιόν να επεκτείνει την ε, σχετική προθεσμία. Τέσσερις από αυτές έχουν μεγαλύτερη πολιτική σημασία γιατί αφορούν ακριβώς ε, την, πώς υπολογίζεται το κεφάλαιο των τραπεζών και έχουν άρα μεγάλη σημασία για την εφαρμογή των οδηγιών ε, και τον αντίκτυπο που θα έχει στο απαιτούμενο κεφάλαιο. Τα δε μέλη μπορούν να δουν ακριβώς ε, το έγγραφο που έχει μοιράσει η Κομισιόν πριν από τη συνεδρίαση και την ομοδότηση της Κομισιόν που επίσης έχετε λάβει. Θα ήθελα τώρα να καλωσορίσω τον ε, Σεμπαστιά ο οποίος είναι τμήματάρχης ε, της αρμόδιας μονάδας και τον Μάρτιν επίσης ο οποίος είναι δημοταρχής ε, του τμήματος τραπεζών και τον Λάσο Φερμπάη, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, στην Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή. Έχετε τον λόγο για 5 λεπτά ο καθένας. Θα ξεκινήσουμε με την Κομισιόν. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε που μας καλέσατε. όπως και το Κοινοβούλιο, θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική δουλειά που γίνεται για τα τεχνικά πρότυπα. Είναι απαραίτητα για να ολοκληρώσουμε το ενίο εγχειρίδιο. Ε, όπως είπατε, Έχουμε εγκρίνει πέντε επιπρόσθετα τεχνικά πρότυπα από την τελευταία φορά και τα τρία τα έχουμε δημοσιεύσει στην ε, επίσημη εφημερίδα και άλλα δύο υπάρχονται ακόμη στη διαδικασία ελέγχου. Άλλα πέντε λοιπόν υπολείπονται που εξετάζονται αυτή τη στιγμή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκ των οποίων τα δύο σχεδίζονται με μεθοδολογίες αξιολόγησης για ε, μοντέλα που χρησιμοποιούν οι τράπεζες ε, για την, ε, τον κίνδυνο στην αγορά και για τον κίνδυνο των δανείων. Όταν ε, ζητείτε δηλαδή αδειοδότηση από τις αρμόδιες αρχές, πώς ε, οι τράπεζες ε, μπορούν να αξιολογήσουν τον κίνδυνο για συγκεκριμένα είδη έκθεσης και έκθεση CVR για τις πρακτικές πρόξη. Και τα πέντε, όπως ε, είπατε, έχουν ήδη εκπονηθεί από την EBA και βρίσκονται σε διαφορετικές φάσεις έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα δύο που, στα οποία αναφερθήκατε και εσείς για τα μοντέλα, την αξιολόγηση κινδύνου, είναι πραγματικά πάρα πολύ περίπλοκα τεχνικά πρότυπα και ε, εσωτερικά χρειάζονται έντονες διαβουλεύσεις και διάλογος με την νομική υπηρεσία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Πρέπει να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι είναι τα καλύτερα δυνατά τα τεχνικά πρότυπα και τα όσο δυνατόν πιο εύληπτα γίνονται για να μπορέσουν να εφαρμόσουν και τράπεζες στη συνέχεια. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ για την έγκριση, για τον κίνδυνο δανείων, για την εσωτερική διαδικασία, δηλαδή εξολόγηση κινδύνου για τις τράπεζες. Ε, έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ και έχουμε προχωρήσει και για δύο άλλα πρότυπα, για το ειδικευμένο ε, ειδικό landing και για την πρώτερη αδειοδότηση, αλλά για το IMA και για τα proxy spreads, για το CVA, έχουμε καθυστέρηση διότι οι πόροι μας ε, έχουν αφιερωθεί ε, στο ε, διαπραγμάτευση του τωρινού πακέτου όπου με μεγάλο κομμάτι είναι ο κίνδυνος αγοράς οπότε οι συνάδελφοι που διοικεύονται στο κίνδυνο της αγοράς είναι πολύ αποσχολημένοι θα προσπαθήσουμε όμως να συνεχίσουμε στο μέτρο του δυνατού τη δουλειά για τα τεχνικά πρότυπα. Πέραν αυτών, ε, εγκρίνουμε τώρα μία τροπολογία στην πράξη εξοδότηση για, ε, για το λόγο ρευστότητα τη κινδυνού. Ε, στα τέλη του περασμένου μήνα καταλήξαμε σε ένα σχέδιο και τώρα ε, εξετάζουμε τα σχόλια που έστειλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς. Ένας από τους λόγους για τους οποίους καθυστερήσαμε την έγκριση ήταν γιατί θέλαμε να περιμένουμε ε, την έγκριση του κανονισμού για τις ε, τιτλοποιήσεις ούτως ώστε στην πράξη κατά εξωσιοδότηση να ενσωματώσουμε τα στοιχεία αυτού του κανονισμού ε, για το LCR, για την κάλυψη της δραστότητας δηλαδή. Ε, ε, κάπου το Μάιο αναμένεται να ολοκληρώσουμε και τα δύο υπολοιπόμενα τεχνικά πρότυπα στα, για τα οποία έχουμε καθυστερήσει. Θα χρειαστεί λίγο περισσότερο χρόνος. Αλλά στην πράξη όλα τα βασικά τεχνικά πρότυπα πολύ σύντομα ε, θα εγκρίνουμε όλα τα τεχνικά πρότυπα λοιπόν, που μας ανέθεσαν η EBA και οι συνομοθέτες. Εσείς από την Επιτροπή θέλετε και δύο το λόγο. Α, είναι κοινή πρόταση, EBA. Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποδίδεται ιδιαίτερη σημασία στην έγκριση των τεχνικών προτύπων. Νομίζω ότι είναι καλό για όλους μας. Ε, με αποτελεσματικό τρόπο και γρήγορα να εγκριθούν αυτά τα πρότυπα, ταυτόχρονα σεβόμενοι το ρόλο κάθε θεσμικού οργάνου. Οποιαδήποτε προσαρμογή της διαδικασίας και βελτίωση της διαδικασίας την καλωσορίζουμε ό,τι μπορείτε να εισηγηθείτε δηλαδή εσείς. Για τα ίδια τα ζητήματα η EBA έχει καταβάλει ιδιαίτερες προσπάθειες ε, κυρίως ε, για τα εσωτερικά μοντέλα για να υπάρχει συνέπεια για την αξιολόγηση του κινδύνου των στοιχείων του ενεργητικού για την ε, μέθοδο αξιολόγησης για την αποτύπωση του κινδύνου γνωρίζετε πόσο σημαντικό είναι για την EBA. Επίσης υπάρχει ένας μικρός αριθμός εντολών που δεν συμπεριλήθησαν τελικά στο CDR4. Περίπου 126 ήταν τα τεχνικά πρότυπα και αντίστοιχα εισάριθμες κατευθυντήριες γραμμές Υπήρξαν ε, καθυστερήσεις κυρίως ε, για, την, ε, για τον κίνδυνο των, της δανειοδότησης επειδή είναι τόσο περίπλοκα και τόσο πολλά τα τεχνικά πρότυπα. Τα υπολοιπόμενα πρότυπα προκύπτουν από πολύ συγκεκριμένες διαβουλεύσεις πρότυπο και προσπαθούμε πάντοτε να ε, αποφεύγουμε την αναβολ, τις αναβολές και τις ε, καθυστερήσεις. Γιατί ε, συμβαίνει όμως παρόλα αυτά αυτό, για να το πω απλά, δύο ειδών είναι οι λόγοι. Για πολλά πρότυπα στο τέλος τη διαδικασία εξακολουθούσαμε να έχουμε πάρα πολλούς ενδιασμούς ε, παρά τι ε, μακροσκελέστατε διαπραγματεύσει ε, και συζητήσει. Δεύτερο είδο λόγων το πακέτο Βασιλείας και η κατεύθυνση που έδωσε η Επιτροπή της Βασιλείας. Νομίζουμε ότι θα δημιουργούσαμε μεγαλύτερη σύγχυση σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητήσουμε τεκμηρίωση, ενώ ακόμη συζητείται το θέμα στην Επιτροπή Βασιλεία. Ζητούνται μεταγενέστερε τροποποιήσει, λοιπόν, παρά το κόστο εφαρμογή για, ε, για τα προ, τεχνικά πρότυπα, εάν τελικά καταφέρουμε ευθυγράμμιση με το πακέτο τη Βασιλεία. Διαδικαστικά, θέλω να σημειώσετε ότι δυνάμεθα να ζητήσουμε περισσότερο χρόνο βάσει του καταστατικού μας για την εκπόνηση τεχνικών προτύπων. Και επιτρέπουμε εμείς πάντοτε ενστάσεις για τις προθέσεις MBA. Και όχι μόνο αυτό, θέλουμε να είναι δημόσιες και διαφανείς ε, οι διαπραγματεύσεις και οι αποφάσεις, ώστε οι νομοθέτες αλλά και το κοινό να γνωρίζουν τι ε, προθέσεις έχει η EBA. Εάν η Επιτροπή μας ε, βάσει του κανονισμού μας δώσει τον επρόσθετο χρόνο, καλώς. Αλλιώς ε, φυσικά προτείνουμε θα προχωρήσουμε και τα τεχνικά πρότυπα. Κατά τα άλλα θα εξακολουθήσουμε να, τη δουλειά που κάνουμε για τα υπόλοιπα τεχνικά πρότυπα. Ευχαριστώ. Ποιοι είναι λοιπόν στην αίθουσα. Ο πρώτος. Ashley Fox. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ε, παρουσίαση που μας κάνατε σήμερα. Εγώ θα ήθελα να εστιάσω το σχόλιά μου στις τροπολογίες όσον αφορά την ε, αναλογία για την κάλυψη της ρευστότητας. Εμείς θα θέλαμε να έχουμε πιο πολύ ευθυγράμμιση ε, γιατί η συμπερίληψη ενός τέτοιου κειμένου δεν καλύπτεται διεθνώς. Το βασικό κριτήριο είναι να μπορεί κανείς να, να, αποσύρει, όπως στην ε, Βασιλεία LCR παράγραφος 53. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος αυτής της διάταξης, δηλαδή να εξασφαλιστούν ε, τα ξένα νομίσματα, ξένα αποθέματα. Αν μπορεί ε, δηλαδή το Ίδρυμα κάθε φορά να αποσύρει, ε, να, μάλλον να κάνει ανάληψη αυτών των αποθεματικών σε οποιαδήποτε φάση ε, στρες θα ήταν αυτό το θετικό στοιχείο. Τώρα με βάση τη Βασιλεία τα, οι, οι κλάδοι αυτοί παίρνουν προτιμησιακό καθεστώς 3% εμείς προτείνουμε να αντικατασταθεί το ESCB, οι Ευρωπαϊκές Συστημικές Ευρωπαϊκές ε, Κεντρικές Τράπεζες με το Eurosystem, γιατί η ERCB περιλαμβάνει και τις ε, τρα, ε, χώρες εκτός της Ένωσης. Αυτό θα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Για το άρθρο 3.11, ο ορισμός του στρες είναι σημαντικό να οριστεί ως μια κατάσταση όπου ίσως υπάρχει και όχι υπάρχει maybe, και όχι there is, ότι το Ίδρυμα δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις δεσπεύσεις του, στις υποχρεώσεις του. Γιατί αυτό δημιουργεί ασυνέπεια με την FDA και περιορίζει τη χρήση των buffers. Θέλουμε να διατηρηθεί ο ορισμός του στρες ως μια περίπτωση όπου δύναται να υπάρχει σημαντικό στρες. Για όλα αυτά μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι αυτέ οι ευθυγραμμίσει με τη Βασιλεία θα γίνουν. τέλο για αυτό το θέμα, στο άρθρο 13, εμεί προτείναμε να εξεταστεί προσεκτικά η ευθυγράμμιση ανάμεσα στην ε, κατοξιδότηση πράξη για, τη ε, για την ε, δέουσα ρευστότητα. Εμεί πιστεύουμε όμω ότι αυτό δεν ισχύει σε σχέση με το τελευταίο. Και όσον αφορά τις ANA, της προσεγγίσης για τον επιχειρησιακό κίνδυνο RTS θα θέλαμε να λειτουργήσουμε σε ένα εναρμονισμένο σύστημα μέσα στο πλαίσιο του ANA. Είναι σημαντικό να αντιμετωπιστούν οι ασυνέπειες καθώς και η μεταβλητότητα, η μη σκόπιμη μεταβλητότητα ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα ENA μέχρι ότου αντικατασταθούν από την τυποποιημένη και μετρημένη προσέγγιση της Βασιλείας. Η καταξιδότηση πράξη δεν αναφέρεται μόνο στα στον επιχειρησιακό κίνδυνο αλλά και στο... στην εφαρμογή ενός συγκεκριμένου ε, πλαισίου για τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει η οθέτηση του από τις μεσές και μεγάλες τράπεζες με στόχο την αποτελεσματική εποπτεία του ΕΝΑ και μια ομαλή μετάβαση των τραπεζών ΕΜΑ στη νέο SMA. Ευχαριστώ. Uh, Finally, we, we have uh, our EPP. Σας ευχαριστώ. Τέλος, ε, ε, βρήκαμε και έναν εισηγητή του ΕΛΚ. Να δώσω το λόγο στον Ότμαρ Κάρα ή θέλετε να μιλήσετε τελευταίος. Mm -hmm. Τώρα θα μιλήσετε. Can do it. Yes. Uh, herzlichen Dank für die Bericht. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση από Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Ταπεζική Αρχή. Θα ήθελα να φέρω κάποια σημεία. Πρώτον, για την επεξεργασία της πράξης κατεξοδότηση για το liquidity coverage ratio. Όλοι γνωρίζουμε πως υπήρξε μία διαβούλευση με τους ενδιαφερόμενους. Ε, υπάρχουν όμως ακόμα δύο ερωτήματα η Κομισιόν θεωρεί σωστό να δούμε και τα στοιχεία ενεργητικού εταιριών ε, προώθησης εξαγωγών τα οποία αξιολογούνται ως ε, εξόχως ε, ρευστά. Θεωρεί ότι θα πρέπει να υπάρξει μια επεξεργασία των κριτήριων ε, όσον αφορά, των κριτηρίων όσον την επαναπεξεργασία του σχετικού κανονισμού. Οπότε φαίνεται οι τιτλοποιήσεις STS ε, ε, έχουν διαμορφωθεί με χειρότερες όρους όσον αφορά την κάλυψη από τρίτες χώρες. Η επόμενη ερώτησή μου αφορεί το RTS για τον επιχειρησιακό κίνδυνο. Τα έχουμε συζητήσει αυτά τον Μάρτιο, Πελιο Μάιο του 2017 και εκεί πέρα μας είπατε ότι η Κομισιόν δηλαδή ότι αυτά θα εγκριθούν τον Μάιο του 2017 και όμως αυτό συνέβη 14 Μαρτίου φέτος. Γιατί αυτή η καθυστέρηση και θα ήθελα να γνωρίζω γιατί ακριβώς ε, προβλέπεται μια προθεσμία εξέτασης ενός μηνός ενώ η Κομισιόν έχει κάνει αρκετές ε, αλλαγές γιατί δεν έχουμε προθεσμία τριών μηνών όπως συνηθίζεται σε αυτές τις περιπτώσεις ε, το τρίτο θέμα αφορά την αξία δανεισμού των στεγαστικών δανείων όπως ξέρουμε έχει παγώσει αυτή η πράξη κατεξιοδότηση καθώς υπάρχει το θέμα των καλυμμένων ομολόγων και των αρνητικών επιπτώσεων στην ευρωπαϊκή αγορά. Και τέλος, μια παρατήρηση για την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής ε, η Κομισιόν θα έπρεπε να της δώσει αυτομάτως ε, να διαβιβάσει αμελητή τον σχετικό κανονισμό. Και βεβαίω θα έπρεπε ακριβώ να υπάρχει μια παράλληλη ταυτόχρονη μετάδοση σε Κομισιόν και Συμβούλιο. Τι άποψη λοιπόν έχει η Κομισιόν εδώ πέρα και γιατί δεν υπήρξε ακριβώς ε, αμέσως ε, αυτή η διαβίβαση. Ποιες βελτιώσεις έχετε να προτείνετε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Γκίγκολτ, θα είμαι πάρα πολύ σύντομος, ε, θα εστιάσω κυρίως σε ζητήματα διαδικαστικά και διοργανικά τα οποία ήδη ετέθησαν και από την εισαγωγή που έγινε οφείλω να πω ότι να το βρίσκω ανησυχητικό ότι ο κανονισμός μας προβλέπει κανονικά την δυνατότητα να απαντήσει η Κομισιόν εντό τριών μηνών και τώρα βλέπουμε ότι κατά κανόνα έχουμε πολύ μεγαλύτερες καθυστερήσεις μας αναφέρατε κάποιους λόγους, αλλά από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένα συστημικό πρόβλημα. Η ίδια Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή χρειάζεται κάποιον χρόνο για να συντάξει τους κανόνες. Εντάξει, αυτό είναι κατανοητό, αλλά φαίνεται ότι μετά και η Κομισιόν ξανά και ξανά χρειάζεται ένα έτος ολόκληρο ή και παραπάνω για να συμφωνήσει σε μια τελική προδιαγραφή. Δεν είχαμε ψηφίσει αυτό. Θα ήθελα λοιπόν ε, να ρωτήσω την Κομισιόν εάν είναι σε θέση τελικά όταν μιλάμε για τεχνικές προδιαγραφές για την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, την ΕΙΟΠΑ και την ΕΣΜΑ να δει τις ε, διαδικασίες της και να διασφαλίσει ότι θα είναι περιορισμένες αυτές οι καθυστερήσεις και να κάνω και μία παρατήρηση. Η εντύπωσή μου είναι ότι ο χρόνος ε, τον οποίο παίρνετε έχει ως αποτέλεσμα μονίμως το ίδιο πράγμα. Να ακούτε τα οργανωμένα συμφέροντα που σας προσεγγίζουν είτε άμεσα είτε εμέσως μέσω των κρετών μελών. Είναι δύσκολο δηλαδή να βρούμε κάποιες τεχνικές προδιαγραφές οι οποίες ε, τελικά κατέληξαν να γίνουν πιο αυστηρές από την Κομισιόν από ό,τι είχαν αρχικά προταθεί. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι πάντα αυτό θέλω. Καμιά φορά μπορεί να υπάρχει αναλογικότητα όντως και λογικό είναι και ενδιαφερόμενοι να κάνουν προτάσεις, αλλά είναι ανησυχητικό εάν ε, μόνο μία κατεύθυνση γνωρίζει η Κομισιόν. Και τουλάχιστον η δική μου εντύπωση αυτή είναι και θα ήθελα να ακούσω κάποιες περιπτώσεις, αν έχετε να μου πείτε, όπου τελικά προχωρήσατε σε ισχυρότερη προστασία των καταναλωτών ως αποτέλεσμα των διαβουλεύσεών σας που τραβάνε πολύ περισσότερο από όσο προβλέπετε. Οπότε, μπορείτε να δεσμευτείτε ότι θα αλλάξετε τις εσωτερικές σας ε, διαδικασίες. Και δεύτερον, αν καθυστερείτε τόσο ε, να ακούτε και τις δύο πλευρές ε, της αγοράς. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε λοιπόν και τεχνικές ερωτήσεις και πιο γενικές. Θα προσθέσω και εγώ μια πιο γενική, γιατί είπατε ότι έχετε την, ε, το τρέχον νομοθετικό πακέτο, το οποίο απαιτεί την χρήση πολλών πόρων αλλά αντιλαμβάνομαι ότι αντιμετωπίζεται πράγματι μια συγκεκριμένη κατάσταση σε σχέση με το RTS που σημαίνει προκλήσεις λόγω και των διαπραγματεύσεων στην Επιτροπή της Βασιλείας. Οπότε, το ερώτημά μου δεν σχετίζεται με τα θέματα μας τόσο όσο με το επόμενο νομοθετικό πακέτο. Προβλέπετε ένα άρθρο που θα μας λέτε να περιμένουμε την Επιτροπή της ε, Βασιλείας. Ποιος άλλος ε, βουλευτής θέλει να μιλήσει και... Όχι. Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τώρα τους πάντες. Ποιος θα ξεκινήσει με την ίδια σειρά. Θα απαντήσω σε κάποια και μετά οι συνάδελφοι στα υπόλοιπα. για το ερώτημα του κυρίου Φόξ. Όλα αυτά τα συζητήσαμε σε σχέση με τις πράξεις κατά και φυσικά τα εξετάζουμε ακόμη. Μπορώ να αγγίθω ποια θα είναι η έκβαση. Μπορώ απλώς να σας πω ότι όλα αυτά τα θέματα τα εξετάζουμε. Μετά. και για την ευθυγράμμιση με τη Βαζιλία και με τον κανονισμό STS. Το ίδιο θα σας απαντήσω. Για τα ερωτήματα του κυρίου Κάρας, για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση, κοιτάζουμε ε, το θέμα ε, της έκθεσης και τις σχέσεις με τις ε, τοπικές αρχές. Θα αφήσω τον συνάδελφο Ματία ε, ε, να απαντήσει στα επόμενα ερωτήματα, αλλά για τα συγκεκριμένα για τη διαδικασία και το, τη διάρκεια τους. Φυσικά έχουμε επίγνωση το ότι μέσα στον κανονισμό προβλέπεται πως τα τεχνικά πρότυπα που υποβάλλονται από την Επιτροπή αναμένεται να έχουν εγκριθεί εντός τριών μηνών. Όταν έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, το κάνουμε. Οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται ε, σε παράβλεψη των καθηκόντων μας ή επειδή κάτι άλλο καλύτερο βρίσκουμε να κάνουμε. Εργαζόμαστε σκληρά για όλα τα τεχνικά πρότυπα που μας στέλνει η EBA. Πολύ καλά γνωρίζουμε πόσο σημαντικά είναι, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Είναι δεδομένοι οι πόροι που έχουμε για να επεξεργαστούμε τα τεχνικά πρότυπα και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο και σας είπα ότι υπάρχουν αντικρουόμενες προτεραιότητες και ε, αυτό ισχύει για, ε, για τους πόρους του ανθρώπινου, το ανθρώπινο δυναμικό που έχουμε. Σας είπα έχουμε το πακέτο για τις τράπεζες, ε, για τον κίνδυνο στην αγορά, έχουμε τις διαπραγματεύσεις στη, Βασιλ, στη Βασιλεία, χρόνος και ε, πόροι, ε, ανθρώπινο δυναμικό χρειάζονται και γι' αυτό είναι απασχολημένοι οι αρμόδιοι. Το ότι καθυστερούμε δεν σημαίνει ότι έχουμε εγκαταλείψει τα τεχνικά πρότυπα. Διακόπτη η κυρία Μπερές. Ο Άσλι Φόξου με ρώτησε για το LCR. Ναι, αλλά είπα ότι όλα αυτά τα ζητήματα τα εξετάζουμε. Απάντησα. Μπερές. Ναι, αλλά δεν μας βοηθάτε. Μα δεν μπορώ να εγγυηθώ τι θα προκύψει από την επεξεργασία και τι όχι. Δεν μπορείτε να μας πείτε, λέει η κυρία Μπερές, τι πήρατε από την EBA. Κάτι να μας πείτε. Αυτό το σκρούτινι που κάνουμε είναι για να ξέρουμε τι γίνεται παρασκηνιακά. Γιατί γι' αυτό ασκείται κριτική. Όταν μας λέτε «Α, ε, το δουλεύουμε και θα σας πούμε όταν τελειώσει», ε, δεν μας ικανοποιεί. Καλά, θα αφήσω τη συνάδελφο να απαντήσει. Εγώ ασχολούμαι με τα γενικόλογα ερωτήματα σε πρώτη φάση. Ε, πρέπει να πω πως ε, δεν είμαι σίγουρος σε ποια τεχνικά πρότυπα αναφέρεστε. Όλα τα τεχνικά πρότυπα ε, για τα οποία εγώ προσωπικά εργάστηκα ή συναδελφοί Ποτέ δεν ήρθαμε σε επαφή με τη βιομηχανία. Ποτέ δεν μου ε, υπαγόρευσαν τι, τι πρέπει να κάνω. Και κανένα δεν αποδυναμώθηκε. Από όσο γνωρίζω εγώ σε σχέση με τις προτάσεις που λάβαμε από την EBA. Καθενίζουμε το κείμενο, διευκρινίζουμε το κείμενο, αλλά δεν αποδυναμώνουμε θα μας βοηθούσατε με συγκεκριμένα παραδείγματα. Δεν ξέρω σε τι αναφέρεστε στο, στις πράξεις κατεξουσιοδότηση ή στα σχέδια που παίρνουμε, αλλά όταν μιλάμε για εφαρμογή τεχνικών προτύπων, ούτε μία περίπτωση δεν μπορώ να σκεφτώ όπου τελικά αποδυναμώσαμε την ε, πρόταση της ε, ΕΜΠΑ. Ε, ίσως ο Λάρς μπορεί να με διορθώσει, αλλά εγώ δεν έχω κάτι στο μυαλό μου. Κάτι πιο γενικό και διαδικαστικό. Αυτή η τρίμηνη διορία. Εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά και το μπορώ να αποκλείσω ότι θα έχουμε και καθυστερήσεις στο μέλλον. Στο παρόν ε, τα τεχνικά πρότυπα σχεδόν εμπρόθεσμα ε, τα δώσαμε. Πάνω από 100 έχουμε πονήσει ήδη και όπως είπε ο και νομίζω πρέπει να το λάβετε υπόψη. Δεν μπορώ να σε εγγύθω ότι δεν θα συντρέξουν λόγια τους οποίους ε, για κάποια τεχνικά πρότυπα θα καθυστερήσουμε σε σχέση με την ε, προτινόμενη, επιβαλλόμενη μάλλον διορία. Θα δώσω το λόγο στο Ματίας για να απαντήσει. Για... Και μετά ε, η Ντελφίν θα δώσει συγκεκριμένα στοιχεία για το LCR. Ματίας, για τον email, κάποια πρόσθετα σχόλια σε σχέση με αυτά που είπε ο Σεμπάστιαν. Να ξέρετε τι σημαίνει όταν παίρνουμε ένα σχέδιο από την ΕΜΠΑ και γιατί υπάρχουν καθυστερήσεις. Όπως είπε ο Σεμπάστιαν, αυτά δεν σχετίζονται με το lobbying που όπως είπατε εσείς. Αλλά ο στόχος είναι να είναι ξεκάθαρες, ε, ε, ξεκάθαρα τα πρότυπα ε, και να υπάρχει σαφήνεια και συνέπεια. Το λάβαμε ναι, το 2015 το σχέδιο και καθυστερήσαμε πάρα πολύ και καταλαβαίνω γιατί είσαστε απογοητευμένοι. Γιατί όμως συνέβη αυτό. ξέρετε ότι καθυστερήσαμε κυρίως ε, λόγω του διαλόγου με την νομική υπηρεσία, γιατί θέλαμε να είναι ξεκάθαρα τα πρότυπα όταν ε, τα εκπονούμε. Γιατί η ίδια η νομική υπηρεσία έχει περιορισμένους, πολύ περιορισμένους πόρους και μετά πρέπει να πάμε στην εμπειρία και να τα ξανασυζητήσουμε. Και για να απαντήσω και στον κύριο Κάρας, γιατί με τον EMA τελικά ε, είχαμε τόσο μεγάλη καθυστέρηση, ε, γι' αυτό. Τώρα, γιατί προτείναμε σκρούτινη μόνο ένα μήνα. Όπως είπε ο κύριο Φόξ, πρόκειται για το στόχο μας για ταχύ εφαρμογή του προτύπου. Επειδή πέρα από τις ε, τροποποιήσεις διατύπωσης δεν υπάρχουν αλλαγές ως προς την ουσία. Θα δείτε τις track changes στο Word, αλλά ε, ε, είναι μόνο η διατύπωση. Γι' αυτό ε, ζητήσαμε αλλαγή του, διαγραμ... του για το σκρούτινι. Σεμπάστιαν, συγγνώμη, κάτι γενικότερο μου ήρθε πάλι. Για τα σχέδια που μα στέλνει η EBA. Πρέπει να το ελέγξω, αλλά πόσο ξέρω. Όταν λαμβάνουμε τα σχέδια από την EBA, Θα στείλουμε σχετικά γρήγορα. Τι σημαίνει γρήγορα, άμεσα, μελετή. Ξέρω εγώ, μία-δύο μέρες. Μπορεί. Ε, κάποιες φορές να μην έγινε αυτό. Και να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε. Αλλά γενικά αυτό ε, κάνουμε συνήθως. Με το που έρχεται το στέλνουμε. Η Δελφίν για το LCR, όπως είπε και ο Σεμπάστιαν, εξετάζουμε τα σχόλια. Δεν έχει εγκριθεί το τελικό κείμενο. Μπορώ παρόλα αυτά να δώσω κάποια στοιχεία για να απαντήσω σε ερωτήσεις των βουλευτών. Για χώρες συμφωνούμε ότι πρέπει να υπάρχει ευθυγράμμιση με τη Βασιλεία για αξιολόγηση μπορεί να είναι προϊόν συμφωνίας ή μπορεί να, και ως λέει να αναγνωριστεί στο LCR σε τοπικό επίπεδο. για τον ε, ορισμό του Trace. Εμείς θέλαμε να ευθυγραμμιστούμε τον ορισμό του CR2 ο ορισμός του στρες, του τεστ ε, κοπόσεως, είναι ότι υπάρχει ε, κίνδυνος και όχι μπορεί να υπάρχει. Ε, το κείμενο SCR e ε, πράξης ε, το ευθυγραμμίζουμε με τον κανονισμό ε, SCR2. E Ο στόχος μας είναι πλήρης ευθυγράμμιση με τον κανονισμό STS, αλλά να διατηρήσουμε και κάποια κριτήρια που σχετίζονται με την ρευστότητα για το LCR. Ε, η σενιόριτη ενός ε, τμήματος ε, δανείου, παραδείγματος χάρη. Δηλαδή πέρα από τα κριτήρια εστίας έχουμε και άλλα που σχετίζονται με την ρευστότητα μέσα στην πράξη κατά εξουσιοδότηση. Κύριε κάρα. Η Επιτροπή δεν θέλει να τροποποιήσει τον ορισμό έτσι και λέει χρησιμοποιούν τον ορισμό της βασιλείας. Ο προτινόμενος ορισμός για να ε, δεχτούμε ότι προέρχεται από ε, agency εξαγωγικών πιστώσεων είναι αυτό στο οποίο βασιζόμαστε και φυσικά είναι αμφιλεγόμενος ο ορισμός ε, του HQLA και της πράξης κατεξοδότητας για το LCR. Πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω λοιπόν. Για να ξέρουμε πόσο ρευστά είναι αυτά τα στοιχεία προτού και αν ε, τελικά αποφασιστεί να τροποποιήσουμε το HQLA. Από την ΕΜΠΑ θέλετε να μας πείτε τίποτα. Ναι, κάποιες ε, παρατηρήσεις. Κύριε Φόξ, νομίζω συμφωνούμε απόλυτα ότι εκτίμηση του EMA θα πρέπει όντως να υιοθετηθεί και αυτό ισχύει και για τις υπόλοιπες τεχνικές προδιαγραφές. Είναι πολύ σημαντικέ για την καθημερινή ε, εποπτεία και πρέπει να υιοθετηθούν. Κύριε Κάρας, σε σχέση με την τους πίνακες της ε, τραπεζικής ε, αρχής, του Υποπτικού Συμβουλίου δηλαδή, ε, θα πρέπει να δείτε ότι από τότε που υιοθετήθηκε αυτή η τιμή προσέγγιση δηλαδή των συστημάτων που χρησιμοποιούν την τιμή αγοράς ε, ε, σημαίνει ότι σημαίνει ότι αξιολογούμε έτσι μόνο ένα κομμάτι της αγοράς, ενώ έχουμε και την ε, αξία των ανυπόθηκων ε, ε, δανείων που θα πρέπει να υπολογιστεί ταυτόχρονα. Θα πρέπει δηλαδή ο νομοθέτης να εξετάσει και τις δύο πρακτικές αλλά και την προσέγγιση που χρησιμοποιεί την αξία της αγοράς, τη τιμή της αγοράς. το Εποπτικό Συμβούλιο θα συνεργαστεί ώστε να βρεθεί συμφωνία ανάμεσα στους ε, νομοθέτες. Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι είναι αρκετά βαριά όλη αυτή η διαδικασία. Ε, η διαδικασία υιοθέτηση, η εξολόγηση των νομικών αλλαγών που προέρχονται από την πλευρά της Κομισιόν φροντίζουμε πολύ να είναι περιορισμένες οι αλλαγές. Σαφώς με τα πιο μακροσκελή κείμενα αυτό ε, καθίσταται ακόμη πιο περίπλοκο. και με την μεθοδολογία αξιολόγησης και τα νομικά κείμενα που φτάνουν τα 100 σελίδες παίρνει πολύ χρόνο αυτό. Και αυτό επιπλέον της αρχικής νομικής ε, ε, εξέτασης του ΕΜΠΑ. Παίρνει πολύ χρόνο ούτω ή άλλως και είναι αυτό πολύ ευπρόσδεκτο. Εντάξει, λέει η κυρία Μπερές. Δεν ξέρω τι θα έλεγε ο πρόεδρος, ο πραγματικός πρόεδρος, αλλά εγώ πρέπει να πω ότι απογοητεύτηκα από αυτόν τον έλεγχο. Πρώτον γιατί λείπαν οι περισσότεροι, αλλά και επειδή δεν μάθαμε και τίποτα καινούριο. Και από ό,τι κατάλαβα, θα πρέπει να ε, αντιμετωπίσουμε ε, μία από τις ανησυχίες από αυτές με τον πρόεδρο της Επιτροπής. Γιατί, γιατί η Επιτροπή οφείλει να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη εφαρμόζουν την νομοθεσία. Το ίδιο ισχύει για την Κομισιόν όταν πρέπει να, να, δράσει σύμφωνα με την κατεξουδότηση πράξη. Οπότε έχουμε πλήρη έλλειψη ευθυγράμμισης και αυτό δεν είναι λογικό. Δεν πήρα και καμιά απάντηση στην ερώτησή μου όσον αφορά την πρόληψη κάποιου ε, πακέτου. Η νομοθεσία λοιπόν θα πρέπει να ακολουθείται και από συγκεκριμένη πρόταση και δεν θα, θα καταλήξουν και θα περιμένουν την Επιτροπή της Βασιλείας να φτάσει στην τη τελική της θέση. Αυτό θα μας επιτρέψει να βάλουμε αυτό το άρθρο εντός παραθέσεων μέχρι ότου αποφασίσει η Επιτροπή της Βασιλείας. Ίσως μπορείτε να μας δώσετε αυτή την απάντηση γραπτός αν θέλετε κάτι τώρα να προσθέσετε σας ακούμε. Εγώ ήθελα να το αφήσω για, τέλος, για το τέλος ως απάντηση. Πιστεύω ότι επί της αρχής, τουλάχιστον όσον αφορά τις προτάσεις της Κομισιόν, εμείς στείνουμε να περιμένουμε την ολοκλήρωση των διεθνών εργασιών πριν να υποβάλουμε τις προτάσεις μας. Σε κάποιο βαθμό λοιπόν, ακόμα και η πρόταση που τώρα διαπραγματευόμαστε που περιλαμβάνει το πλαίσιο για τον κίνδυνο της αγοράς που δεν έχει τελειώσει τελείως στη Βασιλεία με βάση την ίδια αρχή ότι δηλαδή η αρχική μας ε, αντίληψη για το πλαίσιο της μεταρρύθμισης στη Βασιλεία ήταν ότι θα ήταν πολύ πιο περιορισμένο εύρους από ό,τι τελικά ε, ήταν. Και γι' αυτό και προβλέψαμε κατεξοδότηση πράξη ε, για την Κομισιόν ώστε να προσαρμοστεί και να λάβει υπόψη τι αλλαγέ. Τώρα βέβαια η κατάσταση είναι διαφορετική και η προσέγγιση που πρέπει να γίνει τώρα εξετάζεται στο Συμβούλιο και στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά όπως είπα, εν γέννη προτιμάμε να έχουμε ε, στοιχεία που περιλαμβάνονται βασικά από τη στιγμή που πρέπει. Και αν αναφέρεστε στα στοιχεία που συμφωνήθηκαν από την Επιτροπή της Βασιλείας πέρυσι, εμείς επίτηδες δεν το συμπεριλάβαμε στην πρόταση της Επιτροπής για τον κίνδυνο το πιστοτικό και τον επιχειρησιακό, γιατί ακριβώ δεν είχαν συμφωνήσει. Τώρα είναι μια δηλωμένη μας προτίμηση και το έχουμε ήδη πει και στο Κοινοβούλιο ότι προτιμάμε ε, τα θέματα που συνδέονται με τον πιστοτικό κίνδυνο και τον επιχειρησιακό κίνδυνο να μείνουν μαζί κατά κάποιο τρόπο. Να μην προτρέξουμε δηλαδή με κάποια κομμάτια της Συμφωνίας της Βασιλείας τώρα, αλλά να περιμένουμε για ένα ε, δυνητικό μελλοντικό πακέτο. Γιατί κάποιες φορές είναι πολύ δύσκολο να τα προσεγγίζουμε ε, κατά τμήματα γιατί είναι αλληλένδετα πολύ συχνά. Γιατί ε, αν λοιπόν ασχοληθεί μόνο με ένα κομμάτι, μπορεί να έχει επιπτώσει μη αναμενόμενε. Αυτά είναι επιχειρήματα που μπορεί να κατανοήσει ο νομοθέτης, αλλά πιστεύω ότι θα ήταν ε, καλύτερο να ενημερώνεται τακτικά τον νομοθέτη ε, γιατί, πρώτον γιατί δεν ε, ε, λειτουργείται στο χρονοδιάγραμμα που έχει προβλεφθεί και έπειτα για την ε, νομοθεσία που είναι υποσυζήτηση, όπου προφανώς έχετε κάποια γνώμη για το πώς θα πρέπει να προχωρήσει και αυτή θα μπορούσε να είναι μια προστιθέμενη αξία. Τουλάχιστον αυτό είναι το μήνυμα από αυτήν την ανταλλαγή απόψε. Σας ευχαριστώ όλους ε, ε, και όλους όσους έμειναν μέχρι το τέλος αυτές τις συνεδρίες και θα ξαναρχίσουμε αύριο στις 9 και 4 με κοινή συνεδρίαση με την τάξη 3.